Τέσσερις δεν έχουν ψηφίσει. Γιατί... five people who haven't voted. Τώρα πέντε δεν έχουν ψηφίσει. Six people. This is a check. Δεν ψηφίζουμε τίποτα, τσεκ κάνουμε. Δύο συνεχίζουν να μην έχουν ψηφίσει. Mrs. De Kaiser is going to vote with her hands? Right. Then with Mrs. De Kaiser we are okay. We got. You have a card, indeed. Oh, brilliant. Then there's one person who hasn't voted. Λοιπόν, η κυρία Ντεκάιζερ δεν έχει πρόβλημα. Ποιο είναι ο άλλο που δεν έχει ψηφίσει? The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Λοιπόν, πρώτη ψηφοφορία για την απαλλαγή του 2012 Γενικός Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, γνωμοδότηση Γκέρενς Υπάρχει μία τροπολογία για την παράγραφο 6. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας. Κατά. Αποχές. Ωραία, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. The is Πέρας της ψηφοφορίας. Νομίζω ότι είναι ομόφωνη ε, η ψήφος, αλλά κάποιος συνεχίζει να μην έχει ψηφίσει. Κάποιου το μηχάνημα δεν δουλεύει. Λοιπόν, εγκρίνεται η τροπολογία αυτή. Τώρα, για την γνωμοδότηση του συνολότητα, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται αλλά συγγνώμη πρέπει και αυτό να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ What is closed? Πέρας ψηφοφορίας Ομόφωνα περνάει η γνωμοδότηση συγχαρητήρια κύριε Γκέρενς. The second uh, Δεύτερη ψηφοφορία πάλι του κυρίου Γκέρενς για το απαλλαγή 12, 8 και 10 ετά. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τροπολογίε. Ψηφίζουμε την γνωμοδότηση του συνολό. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και εδώ ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση ομόφωνα. Πάλι συγχαρητήρια κύριε Γκόρενς. Η επόμενη γνωμοδότηση είναι δική μου. Εγώ ήμουν ο εισηγητής για το ρόλο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ακίνητης ιδιοκτησίας και τη δημιουργία πλούτου για την εξάλληψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε αναπτυσσόμενες χώρες. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες. Αρχίζουμε με τη συμβαστική τροπολογία Α. Ποιος είναι υπέρ. Hands up, those in favor. Can you count it? No, no, because we, we need to count it, we do it electronically. Let's do this electronically. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και για το θέμα αυτό. Είναι πολύ δύσκολο να μετρήσουμε, λοιπόν, ηλεκτρονικά. Can she indicate? Can she indicate my show? You got your voting card? Take your time. Okay, the vote. Let us vote. The vote is open. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Ψηφίζεται υπέρ. Ωραία. Ε, εν περιπτώσει εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, ωραία, αποχές Εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 37. Υπέρ. Κατά. Αν το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. ψηφίζεται υπέρ, οπότε εγκρίνεται. ...38... ...τροπολογία 38... ...υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...εγκρίνεται... ...τροπολογία... 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 για την παράγραφο 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Πρέπει να το ελέγξουμε λοιπόν. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Amendment 41. Τροπολογία 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Ψήφισαν όλοι παρά παράς ψηφοφορίες Απορρίπτεται. Τροπολογία 42. Block, I, I, could we do block up to 42. Τροπολογία 42. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται φεμ 5 υπέρ κατά κατά από την Επιτροπή Γυναικών. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3. Και θα τη δείτε την προφορική τροπολογία στο τέλος του κειμένου. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 49, υπέρ, Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. Ψηφίσατε. Α, συν δύο υπέρ. Ωραία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51. I did say what is open. Ε, λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για την 51. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά. Ας το δούμε λοιπόν, το ελέγξουμε. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εσείς τι κάνετε, ψηφίστε με ανάταση χειρός. Δεν έχετε καρτούλες, αλλά είστε υπέρ. Πολύ ωραία, δεν πειράζει, απορρίπτεται. Λοιπόν, τροπολογία 54. Η ΣΥΑΡ ζήτησε ψηφοφορία σε τμήματα. Τμήμα πρώτο. Ποιος είναι υπέρ. Πρώτο τμήμα, ε. Κατά. Άρχεται ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίστε. Πέρας. Εσείς είστε υπέρ. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος ψηφίζουμε ηλεκτρονικά υπέρ ε, μάλλον ψηφίστε με συγχωρείτε πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται Amendment 55. Τροπολογία 55. Είστε όλοι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Αποχές. και αυτό θέλει ελέγχο. Ψηφίστε ηλεκτρονικά τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 56 ζητήθηκε από την ECR ε, ψηφοφορία σε τμήματα. Για το πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ελέγξουμε. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τμήμα 2 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός ψηφίστε πέρα αυτής της ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία β του κυρίου Πόγκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Αποχές εγκρίνεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6 τώρα για το αρχικό κείμενο υπέρ κατά δύσκολο. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Τσεκ. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική Συμβαστική... σί, Υπέρ Κατά Έλεγχος Πάντα <laughs> Άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και πάμε στην ψηφοφορία, στην τροπολογία 68, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 69, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 72 σε τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίστε. Ψηφίσατε. Πέρας της ψηφοφορίας. Αγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εβδομήντα έξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές check Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε λοιπόν. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. What is closed. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Από την Επιτροπή Γυναικών, όχι, 7. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Αυτή ήταν η 79, συγγνώμη. Τώρα, η 7 από την Επιτροπή Γυναικών, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική υπαριθμό 5 από τους πράσινους, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Ψηφίσατε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. So, Feb 8 we have to vote on. Yeah. What is, uh... Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Υπέρ κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία D του κυρίου Πόγκα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά τμήματα ε, στην τροπολογία 84 του κυρίου Μίτσελ. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση, άρχεται η ψηφοφορία. What is, Ψήφισαν όλοι, πέρασε ψηφοφορία. Yeah. 86. Απορρίπτεται, 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 16, αρχικό κείμενο υπέρ κατά επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 87. Κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, ε, κατόπιν αιτήματος του ΕΛΚ. Α, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 2, υπέρ, κατά, επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. All voted. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Κατά τμήματα για τη ΦΕΜ 10 από τους πρασίνους. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Άποχες, συγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Άποχες. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Η καταπίπτη 91, φεμ 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Φεμ 3, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 7 των πρασίνων υπέρ. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία για να κάνουμε μια επαλήθευση. Ψήφισαν όλοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τη ΦΕΜ e 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΦΕΜ e 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, τα ψηφίσμα μπλοκ τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ. Κατά. τα Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορία. ψήφισαν όλοι. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία F. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Θέλετε να κάνουμε μια επαλήθευση. Να την επαληθεύσουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση τη ψηφοφορίας. It's carried. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Abstentions. Αποχές. Να κάνουμε μια επελήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. What closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 23. Υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 24 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 25 υπέρ Συγγνώμη, ξέχασα τη D. Υπέρ της D. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφοροκή τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Everyone voted. Ψήφισαν όλοι. Λείπει μια ψήφος, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. block. Ψηφίζουμε μπλοκ τις 27 έως και 33. Μπορούμε να ψηφίσουμε μπλοκ. Όχι. Θα σταματήσουμε στην 32. Ωραία. Unblock. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σχέδιο έκθεσης ως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά. αποχές εγκρίνεται. Να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση όμως. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ωραία. Πέρασε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται λοιπόν το σχέδιο έκθεσης. Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε το σχέδιο ψηφίσματος. Ηλεκτρονικά. είπε ε, άρχεται ψηφοφορία. Those in favor first, do this properly. Those against. Να το κάνουμε σωστά. Υπέρ, κατά. Άρχεται η ψηφοφορία για να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά, λέει ο πρόεδρος τώρα. What is closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία ψηφοφορία για σήμερα είναι η έκθεση της κυρίας Αργεντίνη για την προώθηση της ανάπτυξης μέσω υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των εξωτερικών βιομηχανών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Paragraph 1. Those in favor. 25 υπέρ κατά. Γκρίνεται. Μήπως να κάνουμε κάποιες εν μπλοκ, όλες μαζί. Όχι. Όχι. Τέλος πάντων. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της φορείας. Απορρίπτεται. Τρόπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία, τροπολογία προφορική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμηματική ψηφοφορία που ζήτησαν οι σοσιαλιστές. για την τροπολογία 28. Για το πρώτο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά δεν έχουμε καλύτερα. Έναρξη ψηφοφορίας ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. Για το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται. Να ελέγξουμε λέτε. Όχι. Ας ελέγξουμε. Έναξη ψηφοφορίας για το τρίτο μέρος της 28, ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. λέγει 29. 29. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Νομίζω. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 από το ΕΛΚ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 32. 33. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 39 φιόνα Χολ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι κρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Έναρξη ηλεκτρονικής ψηφορίας. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Ζητώ συγγνώμη, κάποιο πρόβλημα είχε το ηλεκτρονικό σύστημα. Ας επαναλάβουμε την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έναρξη. Ψηφίστε για την τροπολογία 40 παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε. Έναρξη ηλεκτρογικής ψηφορίας. Πέρας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Και εδώ με μια ψηφοδιαφορά. Προφορική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 45 καλύπτεται, 46 έχει αποσυρθεί, 47 τμήματική ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα. Η υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Για το δεύτερο τμήμα. Πρόεδρος, κάτι ρωτά τη γραμματεία. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Ένα λεπτάκι λίγο. Έχουμε ένα τεχνικό θέμα. Προφορική τροπολογία 3. Το δεύτερο τμήμα έχει καταπέσει. Λοιπόν, προφορική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. γκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 52 έχει αποσυρθεί. Για την παράγραφο 24 έχουμε μια τμηματική ψηφοφορία ε, για το πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Όχι. Ζητάτε έλεγχο. Ωραία. Ας ελέγξουμε. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 14 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τρίτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. αποχές. Θα το ελέγξουμε αυτό όμως. Έναρξη ψηφορίας για την 54. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. η ε, προφορική του τροπολογία 4 που βασίζεται στην 55. Προφορική 4 υπέρ. Ναι, ψηφίζουμε για την προφορική τροπολογία 4. Όχι, δεν καταπίπτει αυτή. Η 4 δεν καταπίπτει. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά έναρξη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα. Εγκρίνεται. Πάμε στη 56. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αλλά αυτό θα το ελέγξουμε. Εξήντε Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ ψηφίστε. Εντάξει. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται με μία ψήφο. Και εδώ. 59. Υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται, λέει ο πρόεδρος. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχέ Αποχές. Απορρίπτεται. 62. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Κατά Καταπίπτει 64-62. Ε, συγγνώμη, 65. Υπέρ. Κατά. Ας το ελέγξουμε πάλι αυτό. Ε, έναρξη ψηφορίας για την 65. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται με μία ψήφο δύο φορά πάλι. Που είμαστε τώρα συμβιβαστική 3. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Μου φαίνεται ότι απορρίπτεται. Μήπως να το ελέγξουμε όμως. Έναρξη ψηφορίας ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφορίας. Και απορρίπτεται. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε για την Τροπολογία 66. Υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. 66. Ψήφισαν όλοι. Πέρα ψηφορίας. Με μία ψηφοδιαφορά απορρίπτεται μήπως να κάνουμε ψηφοφορίες εν μπλοκ. Από το 67 μέχρι το 74 ίσως θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε όλες μαζί. 67 μέχρι την 74. Ποιοι είναι υπέρ σε αυτό το μπλοκ. Κατά. Απορρίπτονται. 75 είναι με την 74, πρέπει ε, προφορική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. citations. Από την 1 μέχρι τη συμβιβαστική 1 στον κατάλογο ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένη και τη συμβιβαστική 1, ομού, από την 1 μέχρι την. Ναι, υπέρ. Κατά. Αποχέ. εγκρίνατε. Επομένω, ε, τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ, υπέρ. κατά ας ελέγξουμε έναρξη ψηφοφορίας ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. Τροπολογία 13 υπέρ Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Ωραία, πέρα ψηφορία. Απορρίπτεται με μία ψηφοδιαφορά. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 5, να τεθεί σε ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, παρακαλώ, εκτός μικροφώνου σχόλιο. Εγκρίνεται η 15. 16, παρακαλώ σηκώνετε ψηλά τα χέρια σας. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 9 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρόπο λέγει 21 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μία ψηφοδίαφορα. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Κοίτα να δεις. Ας κάνουμε έναν έλεγχο και εδώ. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφορίας. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην έκθεση λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το σύνολο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Πρώτα απ' όλα μάλλον διανάτες χειρός υπέρ. Καλά, ας ελέγξουμε καλύτερα. Ας κάνουμε την τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, αρκετά μεγάλη διαφορά. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια κυρία Σαρτζεντίνη. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, ας ε, ξανά συγκεντρωθούμε για να συνεχίσουμε. On a subject that, uh, Ανταλλαγή απόψεων ενδιαφέρουσα για ένα θέμα το οποίο ποτέ δεν το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ στην Επιτροπή μας. Εννοώ την ανθρωπιστική δράση μη κρατικών ενόπλων δυνάμεων όμως με σκοπό την προστασία των ε, παιδιών. Η κυρία Σαρτζεντίνη είναι η συγγήτρια ε, για αυτό το πολύ καινούριο θέμα. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Αύριο είναι η διεθνή ημέρα κατά της στράτευσης στρα... παιδιών και προτείνουμε οι πράσινοι να, στην Επιτροπή αυτή να εκδώσει ε, σύσταση προς το Συμβούλιο για το θέμα αυτό και σχετικά με τη δράση μη κρατικών δυνάμεων. Lord's Resistance Army παραδείγματος χάρη όπου χρησιμοποιούν τα παιδιά σαν κατασκόπους, σαν στρατιώτους σαν ε, αγγελιοφόρους και τα λοιπά. Πώς μπορούμε λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με μη κρατικέ δυνάμεις, ένοπλες όμως, ε, και να τους πείσουμε να μην χρησιμοποιούν τα παιδιά σε μια σύραξη. Είναι ένα θέμα που συζητήθηκε από μια πολύ εξειδικευμένη οργάνωση, Geneva Call, που υποστηρίχθηκε από το καντόνι της Γενέβης στην Ελβετία και από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και η οργάνωση αυτή προσπάθησε να έρθει σε επαφή με, αυτούς τους, με αυτές τις μη κρατικέ δυνάμεις για να τις πείσει να μην χρησιμοποιούν τα παιδιά με, οποιοδήποτε λόγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα Κάφριν Άστον, είναι υπέρ της προσπάθειας αυτής γιατί θέλουμε πραγματικά όλοι μας να απαγορεύεται η χρησιμοποίηση παιδιών σε ένοπλες σειράξεις για οποιοδήποτε λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαρτζεντίνη, λέει ο πρόεδρος. Δεν ξέρω αν οι συνάδελφοι, κάποιος συνάδελφος θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ο κύριος Κορτές Λάστρα. Ευχαριστώ. Μιλάω εξ ονόματος του σκιώδη της εισηγητή των σοσιαλιστών, τον κύριο Νόλσεν και θα ήθελε να δείξει και ότι η ομάδα μας ευαισθητοποιείται για το θέμα αυτό και επίσης να επισημάνουμε ότι όλες οι πρωτοβουλίες που προτείνονται στην έκθεση αυτή, κυρίως το θέμα της προστασίας των παιδιών ε, σε ένοπλες σειράξεις ε, και αυτός ο ειδικό εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά να αναγνωρίσουμε, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε και το ρόλο του διαδραματίζουν τα Ηνωμένα Έθνη στην προστασία αυτών των παιδιών, να αναγνωρίσουμε και τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει πάντα να προέχει αυτός ο στόχος για να προστατεύσουμε ανήλικα παιδιά κάτω των 18 ετών. Ε, συμφωνούμε με τα όσα προτείνει η κυρία Σαρχεντίνη στην εκθεσή τη και θα προτείνουμε κάποιες τροπολογίες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πολύ. Uh, thank you very much. Και εγώ ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Άλλος που θα ήθελε το λόγο. Μαρία Λέντ. Ευχαριστώ. Λέγομαι Μαρία Λένσου, ε, εργάζομαι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Κομισιόν χαιρετίζει τη σύσταση αυτή γιατί πραγματικά ε, σε ένοπλες ε, σειράξεις ε, πολλές φορές συμμετέχουν μη κρατικές ενόπλες δυνάμεις ε, οι οποίες χρησιμοποιούν παιδιά. Εμείς προσπαθούμε να ε, επέμβουμε η ΕΚΟ παραδείγματος χάρη, η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ αυτή τη στιγμή ασχολείται με το θέμα της ανθρωπιστικής δράσης ε, και με, σε σχέση με κρατικές και με μη κρατικές δυνάμεις. Υπάρχουν ε, ε διάφορες δράσεις που έχουν ήδη ε, αποφασιστεί και που σχετίζονται με χώρες όπως το Ιράκ, το, η Κολομβία κτλ. Υπάρχει ε, επίσης ένα πρόγραμμα της Γενέβης στο Σουδάν Παλιότερα η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ υποστήριξε άλλο ένα πρόγραμμα της Geneva Call όπου προέβλεπε κατάρτιση ε, για ε, διάφορους συμμετέχοντες στην Ταϊλάνδη και κάτι αντίστοιχο στη Σομαλία. Σε γενικές γραμμές η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ αναφέρεται, ε, διαθέτει 12% του προπολογισμού της για την προστασία των παιδιών. 800.000 ε, ευρώ πέρσι δώσαμε για οργανώσεις προστασίας παιδιών και όμως ε, είναι ε, χρειάζονται παραπάνω χρήματα διότι υπάρχουν πολύ περισσότερα παιδιά που πρέπει να προστατεύσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Δεν ξέρω αν η κυρία Σαρτζεντίνη θέλει να κάνει κάποιες τελικές παρατηρήσεις μετά από αυτά που ακούστηκαν. Ναι θα είμαι πολύ σύντομη. Αν κατά τύχη κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να βελτιώσει την πρότασή μας δεν λέω να την διορθώσει λέω να την βελτιώσει η, διορία είναι έχει χρόνο να το κάνει μέχρι αύριο στις 5 η ώρα το απόγευμα ε, αν θέλετε λοιπόν να προτείνετε κάποιες βελτιώσεις κάντε το μέχρι αύριο στις 5 η ώρα και πιστεύουμε ότι με τη σύσταση αυτή το Ευρωπαϊκό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτεί φόρο τιμής στη σημερινή Διεθνή ημέρα κατά των παιδιών στρατιωτών και η ζητούμε από την Κάθριν Άστον να βοηθήσει ε, σε σχέση με τις μικρατικές δυνάμεις ε, για την προστασία των παιδιών. Βερονίκ, ναι, θέλω, πήρα το λόγο για να πω στην κυρία Σαρτζεντίνη ότι στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ψηφίσαμε ε, ένα ψήφιμα κατά των βασανιστήριων ιδιαίτερα για τα βασανιστήρια των παιδιών και το θέμα των παιδιών στρατιωτών αναφέρεται και σε εκείνη εκεί την έκθεση κατά των βασανιστήριων. Δεν πειράζει, είναι καλό αυτό, το, το ξαναλέμε, το τονίζουμε και πραγματικά όσο περισσότερο επιμένουμε σε διαφορετικά επίπεδα και σε διαφορετικά βήματα τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ λέει ο πρόεδρος. Προχωρούμε τώρα. Yes, um, Judith mentioned it. Um, I'm supposed to tell you formally Πρέπει να σας πω επισήμως μου λένε ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι στις 12 Φεβρουαρίου αύριο. <coughs> στις 5 η ώρα και η ψηφοφορία θα γίνει στις 3 Μαρτίου, στην επόμενη συνάντησή μας. Προχωρούμε τώρα στο σημείο 19. Ενδιαφέρον και αυτό, Um, θα ήθελα λοιπόν αγαπητοί συναδελφοί να καλωσορίσουμε τον εκπρόσωπο των βιβλιοθηκών χωρίς σύνορα ο οποίος θα μοιραστεί μαζί μας την ευρύτατη εμπειρία που έχει σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας σε πάνω από 20 χώρες παγκοσμίως. Ε, Είμαι βέβαιος ότι αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα κινητοποιήσει τους ευρωβουλευτές για να υποστηρίξουν το κατεπήγον ζήτημα της ανάγνωσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, κάτοχοι βραβείων Νόμπελ, συγγραφείς και εμπειρογνώμονες έχουν ασχοληθεί με το θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από τον ε, αρμόδιο, να, τον κύριο Λάκλαλ, να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αγαπητούς ευρωβουλευτές. Η Βιβλιοθήκη Χωρίς Σύνορε είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση που δημιουργήθηκε από ένα Γάλλο ιστορικό, τον κύριο Νίλ Πατρίκ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι εδώ αυτή τη στιγμή, βρίσκεται μεταξύ Γαλλίας και Ηνωμένων Πολιτειών, ζητά συγγνώμη λοιπόν για την απουσία του. Εγώ συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο των Βιβλιοθηκών Χωρίς Σύνορα και ε, ασχολούμαι με κάποιες δραστηριότητες ε, και είμαι συνεργάτης του Γενικού Διευθυντή. Θα ήθελα να σας κάνω μια σύντομη γενική παρουσίαση των Βιβλιοθηκών Χωρίς Σύνορα και από εκεί και πέρα να σας παρουσιάσω δύο συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία επικεντρώνονται πολύ ε, στις δραστηριότητές μας αυτή τη στιγμή. Εγώ ήμουν πρέσβη τη Γαλλία στην Αιτή όταν ξεκίνησαν οι βιβλιοθήκε χωρί σύνορα και οι βιβλιοθήκε χωρί σύνορα έκαναν την πρώτη του ε, αποστολή στην Αιτή. Τότε ήθελαν απλώ να διανύμουν βιβλία. 20.000 βιβλία απεστάλησαν στην Αιτή ε, και πωλήθηκαν με κόστο ευρώ το βιβλίο. Στη Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες, νομίζω, πολλές φορές όταν ε, δορίζει κάποιος βιβλία σε χώρες του τρίτου χώρου, του τρίτου κόσμου δάνουμε τα πλεονέσματα τα οποία συλλέγουμε και πολλές φορές όταν φτάνουν αυτά τα βιβλία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, δεν μπορούν να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες και επομένω δεν ξέρω και αν είναι αποτελεσματική η δωρεά αυτή. Οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα δίνουν βιβλία χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή με τους ε, αποστολείς, ε, ε, συζητούν με βιβλιοθηκονόμους και πολλές φορές τα βιβλία επιλέγονται με βάση τις ανάγκες στον τελικό προορισμό. Έχουν έρθει σε επαφή με πολύ μεγάλους εκδοτικούς οίκους και μεγάλες γαλλικές βιβλιοθήκες, όπως επίσης και βιβλιοθήκες ε, άλλων γειτονικών χωρών και διαθέτει ένα κατάλογο 300.000 βιβλίων. Κάποια από αυτά τα βιβλία διατίθεται δωρεάν και κάποια άλλα με μειωμένη τιμή και προσπαθούμε να ε, καλύψουμε τις πραγματικές ανάγκες και να κάνουμε μια ευφυή και λογική διανομή. Οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα ε, πρόσθεσαν στις αρχικές του δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα την κατάρτιση βιβλιοθηκονόμων ή και ανθρώπων που διαχειρίζονται βιβλιοθήκες και ε, στις αρχές του 2010 είχαμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός ε, το οποίο ε, ε, οδήγησε σε εκτοπισμούς ανθρώπων και οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα ε, που ήταν ήδη επιτόπου στην ΑΕΤ προσπάθησαν να δημιουργήσουν χώρους όπου, που θα λειτουργήσουν ως βιβλιοθήκες για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν στερηθεί τα πάντα. έτσι ώστε να έχουμε μικρά πολιτιστικά κέντρα για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες αλλά τα κέντρα αυτά γνώρισαν μεγάλη επιτυχία και επέτρεψαν στα παιδιά στην ΑΕΤ να έχουν έχουν έστω κάποια σχολική δραστηριότητα χάρη στα βιβλία τα οποία τους διατέθηκαν. Οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα ε, προσπάθησε μέσω των δραστηριοτήτων της ε, να αυξήσει ε, τα όσα έκανε και αυτή τη στιγμή δεν είναι απλώς μια ένωση ε, πολιτιστικού χαρακτήρα αλλά μια κυβερνητική οργάνωση που βοηθά την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη. Οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα θέλουν να δίνουν στις πιο ευάλωτες ομάδες ανθρώπων ε, μέσα για να μπορέσουν να γνωρίσουν τον κόσμο, να μπορέσουν να αλλάξουν και να αντιληφθούν ότι η πρόσβαση στην ε, μόρφωση, στην παιδεία, στον πολιτισμό είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη του ανθρώπου και της κοινωνίας και για να μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους της χιλιετίας όχι μόνο στον τομέα της παιδείας αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς, κυρίως στον τομέα της υγείας αλλά και σε πολλούς άλλους. Αυτό μας οδήγησε στο ε, να σκεφτούμε την όλη έννοια της βιβλιοθήκης εκ νέου και ε, ξέρουμε ότι η βιβλιοθήκη προσφέρει περιεχόμενο, προσαρμόζεται στις ανάγκες του καθενός και στις φτωχότερες χώρες, ε, διότι δεν θέλουμε απλώς ε, να ε, μάθουμε στον κόσμο να διαβάζει βιβλία, αλλά να καταπολεμήσουμε, να και αυτή την ψηφιακή εισβολή και γι' αυτό ακριβώς οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα προσαρμόζουν στα γαλλικά τα παιδαγωγικά μέσα της ε, Γαλλικής Ακαδημίας και αυτό προσφέρει και συγκεκριμένο περιεχόμενο για τους ε, γαλλόφωνους χρήστες και αυτό το περιεχόμενο δεν διατίθεται μόνο σε φοιτητές, σε καθηγητές και σε ερευνητές όπως γίνεται συνήθως, αλλά και σε όλους όσους θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν για τα θέματα αυτά, ιατροί, νομικοί, γιατί όχι και επιχειρηματίες, τις χώρες τις οποίες ε, δεν υπάρχει ευκολία σύνδεσης διαδικτύου. Ε, υπάρχουν προβλήματα στο να είναι κάποιος συνδεδεμένος ή να μπορεί να χρησιμοποιήσει υπολογιστή. Οι βιβλιοθήκες λοιπόν χωρίς σύνορα πρέπει πολλές φορές να μεταβούν στις πρωτεύουσες κάποιων χωρών για να μπορέσουν να φορτίσουν τους υπολογιστές τους, για να μπορέσουν να έχουν επικυροποιημένους ε, ε, υπολογιστές χώρες οι οποίες στερούνται τα πάντα. Πέραν όμως από τη συνήθη λειτουργία της βιβλιοθήκης, η οποία εμπλουτίζεται και από την σύγχρονη τεχνολογία, οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα θεωρούν ότι οι βιβλιοθήκες είναι ένας χώρος συνάντησης ανθρώπων για να μπορέσουμε να ε, δημιουργήσουμε γνώσεις, ε, να μπορέσουμε να απτύξουμε κριτικό πνεύμα και δημοκρατία. Ε, υπάρχουν μεγάλες ανισότητες ε, που μπορεί να είναι λόγω της φτώχειας για παράδειγμα σε χώρες όπως ο Νίγηρας, ε, ε, θεομηνίες όπως ε, στην Αϊτή ε, ή πόλεμοι όπως στη Συρία και οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα προσπαθούν να μάθουν στους ανθρώπους να πάρουν κάποιο χρόνο για να μάθουν να διαβάζουν, να μορφώνονται και να συνεργάζονται. Γι' αυτό ακριβώ υποστηρίζουμε όλες τις βιβλιοθήκες, σχολικές, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, δημόσιες βιβλιοθήκες, αλλά και κινητές βιβλιοθήκες, ε, βιβλιοθήκες κάτω από κάποια σκηνή ή και ε, κινητές βιβλιοθήκες που μπορούν να μεταφερθούν κατεπηγόντως κάπου αλλού, ε, όπου χρειαστεί, εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα προσπαθούν να καταπολεμήσουν και αυτό το ψηφιακό κατακαιρματισμό και προσπαθούν να προσφέρουν κάποια μέσα τα οποία διατίθεται και χωρίς σύνδεση διαδικτύου. Όλες αυτές οι δράσεις ε, μας οδήγησαν να πάμε λίγο περαιτέρα και οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα πλέον συμμετέχουν άμεσα στην οικονομική ανάπτυξη κάποιων χωρών, για παράδειγμα ε, υποστηρίζοντας ε, ε, δίκτυα διανομής βιβλίων σε τοπικό επίπεδο, το να μπορούν να διαθέτουν οι βιβλιοθήκες βιβλιοθηκονόμους, ε, ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να μάθουν και πώς ε, ε, λειτουργούν οι πολιτικές δανεισμού και απόκτησης βιβλίων, καθώς επίσης και οικονομικά, ανθρωπιστικά συστήματα τα οποία επιτρέπουν να συνεχίζονται και να προωθείται η πολιτιστική βιομηχανία οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα μπορούν πλέον να ε, δημιουργήσουν ε, και πολιτιστικές ε, πολύ μικρές επιχειρήσεις που οι οποίες μπορούν να ζητήσουν χρηματοδότηση. Όπως σας είπα οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα δημιουργήθηκαν το 2007 και μέχρι σήμερα έχουν 28 υπαλλήλους, 300 εθελοντές παγκοσμίως, 70% στηρίζονται σε ιδιωτική χρηματοδότηση και 30% σε δημόσια χρηματοδότηση, όπως για παράδειγμα χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τέσσερα δίκτυα ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Ελβετία και στο Βέλγιο που μπορούν να λάβουν κονδύλια, καθώς επίσης ε, ε, χάρη σε αυτά τα μέσα οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα προσπαθούν να αναπτύξουν αυτή τη διπλή πολιτική, δηλαδή να αντιμετωπίζουν κατεπίγουσες καταστάσεις, αλλά ταυτόχρονα να προωθούν και να προάγουν τον πολιτισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Λασάλ. Σας ευχαριστώ. Όπως είπε και ο Χριστιαν πριν από λίγο και όπως εξάλλου μας είχε προτείνει και η κυρία Ευαζολή όταν συναντηθήκαμε στην ε, στη, διεθνή διάσκεψη για τη σημασία της ανάγνωσης τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει σημασία να προωθήσουμε την ανάπτυξη και προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνουμε το πρόγραμμα Ideas Box προσπαθώντας να επέμβουμε σε καταστάσεις επίγουσας ανάγκης στο πεδίο. Θα ήθελα κάπως να σας εξηγήσω πώς ε, ήρθαμε σε αυτόν τον τομέα, γιατί όπως γνωρίζετε εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που ασχολούμαστε με τις ανθρωπιστικές καταστροφές, ασχολούμαστε με πιο μακροπρόθεσμους στόχους. Ωστόσο μας ζήτησαν οι εταίροι, οι εταίροι μας, οι ε, οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόμασταν να επέμβουμε σε καταστάσεις, σε περιοχές τις οποίες υπήρχαν καταστροφές ε, ε, επίγοντος χαρακτήρα και να δημιουργήσουμε βιβλιοθήκες, κινητές βιβλιοθήκες τις οποίες ο κόσμος θα είχε πρόσβαση στην πληροφορία και θα είχε τη δυνατότητα να έρθει και να διαβάζει βιβλία. Και συνέβη κάτι το οποίο δεν περιστρέφει δεν περιμέναμε ότι αυτές οι κινητές βιβλιοθήκες γίνανε πραγματικά σημεία μια συνάντηση. Δηλαδή ήταν ένας τόπος στον οποίο μπορούσαν οι άνθρωποι να ε, ε, συναντηθούν με ασφάλεια. Ήταν ε, ένα safe space όπως λέγεται στην γλώσσα των ανθρωπιστικών αποστολών. Ήταν ένας χώρος στον οποίο θα μπορούσαν να συναντηθούν υπό αυτές τις ασφαλείς συνθήκες και για παράδειγμα οι γιατροί χωρί σύνορα μας επισκέφθηκαν σε μια τέτοιου είδους βιβλιοθήκη και μας είπαν εξαιρετικά σημαντικό αυτό που κάνετε γιατί η ανθρωπότητά μας το βασίζεται στην ε, ικανότητα μας, τη δυνατότητά μας να επικοινωνούμε, να γράφουμε, να μιλάμε. Και αυτή η ανάγκη είναι πραγματικά θεμελιώδης και την καλύπτουμε με αυτούς τους, ε, τις δράσεις. Έτσι λοιπόν η Διεθνής Εκστρατεία The Urgency of Reading, η επίγουσα ανάγκη της ανάγνωσης, είναι μια εκστρατεία η οποία τυχαίνει ε, ευρύτατης υποστήριξης όπως είπατε και εσείς. Μια εκστρατεία που μας έκανε να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την ανάγκη. Η Επιτροπή για τους Πρόσφυγες και ο σχεδιαστής Σταρκ ε, μας ε, δημιούργησε αυτό το, το, το, την κατασκευή που βλέπετε βασικά, που στηρίζεται σε δύο παλέτε και την βλέπετε στην οθόνη σα, η οποία στην πραγματικότητα είναι, είναι πολύ μια πολύ εύκολη μικρή φορητή βιβλιοθήκη, στην οποία μπορεί κάποιο να καθίσει και να έχει ε, πρόσβαση στο ίντερνετ μέσω ταμπλέτα, μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν κατάλογο πάνω από 5.000 τίτλων, έχει επίση ένα σινεμά, μπορεί κανεί να δει ταινίε μέσω μια ε, με οθόνη τηλεόραση και επίση δίνουμε τη δυνατότητα έκφρασης, δημιουργικής έκφρασης στον πληθυσμό που έχει πληγεί από την επίγουσα καταστροφή. Το, το, πιο ενδιαφέρον για μένα αυτή τη κατασκευή είναι το πόσο φορητή είναι και το πόσο εύκολο είναι να δημιουργηθεί γρήγορα ένας τέτοιος τόπος ασφαλής και φυσιολογικός σε μια κατάσταση επίγουσης ανάγκης. Σας δίνω τώρα μια κάποια εικόνα των παρεμβάσεών μας και που βρισκόμαστε σήμερα και που πρόκειται να, ε, ε, να πάμε. Στα πρώτα Ideas Box τα χρησιμοποίησαμε, τα δημιουργήσαμε στο, στη Ρουάντα το καλοκαίρι του 2014. Ε, μάλλον σκοπεύουμε να. Ε, πάμε εκεί. Ε, το Μπουρούντι και στην Μέση θα ήθελα να σα δώσω μια εικόνα επίση του κόστους αυτού του Ideas Box, γιατί πολύ συχνά λέμε ότι οι βασικές ανάγκες είναι πιο σημαντικές και όλα αυτά τα πολιτιστικά αγαθά έρχονται δεύτερα. Όμως, με μια κατασκευή σαν αυτή που έχουμε φτιάξει, στην πραγματικότητα χρειάζονται μόνο 15 δολάρια ανά άτομο που θα αποφεληθεί, το οποίο θα ότι είναι εξαιρετικά ε, καλή κόστου ε, κόστους-οφέλους δεδομένου του πόσο άνθρωποι τελικά αφορούνται από αυτή την πρόσβαση στην πληροφορία. Η πρόσβαση στην πληροφορία είναι πολύ πιο ακριβή. Η ιδέα λοιπόν είναι να προφυλάξουμε τον πληθυσμό από αυτό το χάσμα, από αυτή την, την πλήρη, από, ε, από το να αποκοπεί πλήρως από την πρόσβαση στην πληροφορία έτσι ώστε, γιατί αυτό δημιουργεί ε, τεράστια προβλήματα, τεράστια προβλήματα στην εκπαίδευση, στο, στη, στην ψυχολογική κατάσταση του πληθυσμού, το γεγονός ότι αποκόπτονται ξαφνικά από ολόκληρο τον κόσμο και από το τι συμβαίνει και από ε, ο, τις συνηθισμένες τους ε, δραστηριότητες και μπορούν ε, με αυτό τον τρόπο να συνεχίσουν να βρίσκονται σε μια κατάσταση πιο συνηθισμένη το Ideas Box λοιπόν, μακροπρόθεσμα και εμέσως, βοηθάει και στην οικονομική ανάπτυξη. Σκοπεύουμε να πάμε στην IT, στη Φιλιππίνες, στο Κεντρική Αφρική, στη Συρία, στο Λίβανο, να επέμβουμε οπουδήποτε υπάρχουν τέτοιες επίγουσες ανθρωπιστικές καταστροφές. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μόνο 10 λεπτά στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό, γιατί έχουμε και άλλα ε, δύσκολα ζητήματα μετά. Έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομο θα είμαι. Δεν γνώριζα καν την ύπαρξη αυτή τη πρωτοβουλία, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχω μια απλή ερώτηση που σίγουρα θα την έχετε σκεφτεί. υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με προβλήματα όρασης και το 85% των ατόμων με προβλήματα όρασης βρίσκονται στην Αφρική. Επομένως είναι πολύ περισσότεροι στην Αφρική από ότι στην Ευρώπη. Επομένως έχετε αυτή την ε, πρωτοβουλία η οποία είναι πράγματι αξιέπαινη, αλλά πώς αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα με τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία σας, έχω εντυπωσιαστεί. Βρήκα επίσης και την φωτογραφία του Στέφαν Χέρσελ, ο οποίος ήταν ένας από φίλους μου και χάρηκα που το είδα αυτό. Όταν επισκέφθηκα τη Συρία, διαπίστωσα ότι η UNICEF βρισκόταν στη Δαμασκό αλλά το μεγάλο πρόβλημα στη Συρία είναι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι και τα 3 εκατομμύρια παιδιών που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο εδώ και τρία χρόνια. Μιας και αναφερθήκατε λοιπόν στη Συρία, είπατε επίσης ε, για την Ιορδανία και για το Λίβανο, σκέφτεστε λοιπόν να πάτε εκεί συνεργαζόμενοι και μέσω των διεθνών οργανισμών που βρίσκονται ήδη στο πεδίο δηλαδή των οργανώσεων που ήδη βρίσκονται επί τόπου και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ε, ανυπαρξίας εκπαιδευτικού συστήματος, τα πολιτιστικά προβλήματα κτλ. Το, έχετε εντάξει αυτό στο σχεδιασμό σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ έχω εντυπωσιαστεί και το ε, βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, δεν γνώριζα την πρωτοβουλία σας πιο πριν. Μια ερώτηση μου ήρθε. Έχει, σας έχει φανεί αναγκαίο να κάνετε κάποιο είδους λογοκρισία ή εν πάση περιπτώσει επιλογή των βιβλίων στα οποία ε, τα δίνεται πρόσβαση, για παράδειγμα θρησκευτικά βιβλία. Γιατί αυτά μπορούν να δημιουργήσουν εντάσεις ή προβλήματα ή διχογνωμίες. Ε, επιλέγετε με κάποιο κριτήριο τα βιβλία στα οποία δίνετε πρόσβαση. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος εκτός μικροφώνου. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πρώτη φορά ακούω για αυτή την πρωτοβουλία και πολύ ενδιαφέρουσα τη βρίσκω. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να υποστηρίζει πρωτοβουλίες ε, τέτοιου τύπου, όπως γνωρίζετε το 2012 το βραβείο Νόμπελ ε, ειρήνης ε, δόθηκε στο πρόγραμμα Children for Peace. Εμείς Χρηματοδοτήσαμε προγράμματα το επευθύνονται σε 28.000 παιδιά τα οποία έχουν ε, πληγεί από τον πόλεμο. Έχουμε αυξήσει την χρηματοδότηση το 2013 σε 4 εκατομμύρια και θα ε, βοηθήσει ακόμα περισσότερα παιδιά. Επομένως το πρόγραμμά σας, η πρωτοβουλία σας μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πριν να δώσω το λόγο στους ομιλητές, να υπενθυμίσω ότι όταν χρειάστηκε να βοηθηθούν πάνω από 300.000 άτομα που ήταν εσωτερικά εκτοπισμένοι, είχαν δημιουργήσει ε, κινητά σχολεία στους καταβλισμούς. Επομένως θεωρώ ότι αυτό που κάνετε είναι θαυμάσιο και θα είχε κάποιο νόημα να ε, εξετάσετε την πιθανότητα να παρέμβετε και σε άλλες χώρες πέρα από τις Αφρικανικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κάποιες πρώτες απαντήσεις να δώσω. Ναι, Όντως οι άνθρωποι που έχουν προβλήματα όρασης μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και ασχολούμεθα με αυτούς την IT παραδείγματο χάρη έχουμε μια ηχητική, ακουστική βιβλιοθήκη για τους, ε, προβλ, για τους ανθρώπους που έχουν ε, τέτοια προβλήματα ερχόμαστε σε επαφή με τους ε, δημιουργούς που φτιάχνουν μουσική και ε, ακουστικά βιβλία. Επίσης και το Ideas Box. Εκεί πραγματικά θα μπορούσαμε να μαγνητοφωνήσουμε ραδιόφωνο, έχει υπάρχουν μικρόφωνα, οπότε θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα, για αυτό που είπατε για τη Συρία, όντως είναι πολύ σοβαρό σοβαρή η ερώτηση αυτή τι μπορούμε να κάνουμε στη Συρία αυτή τη στιγμή αρχίσαμε να δουλεύουμε στην Ιορδανία και στο Λιβα... Λίβανο και το 2014 θα αρχίσουμε την αναδίπλωση. Αν θέλετε τον uh, Ideas Box εκεί φορητών κουτιών που μπορούν να μεταφέρουν τα κινηθούν εύκολα και να πάνε να βρουν αν θέλετε μετανάστες όχι που είναι μέσα σε ε, καταβλισμούς αλλά μέσα στις πόλεις προσπαθά μοιραία θα εκτιμήσουμε θα αξιολογήσουμε τι θα γίνει εκεί για να δούμε πως μπορούμε να προχωρήσουμε το 2015 θα φροντίσουμε να διαδώσουμε ακόμη περισσότερο το Ideas Box και βεβαίως ελπίζουμε να υπάρχει κάποια στήριξη αρκετή ούτως ώστε να μπορέσουμε να πάμε και πέρα από την Ιορδανία και το Λίβανο και στη Συρία. Κοιτάξτε τώρα, ε, εδώ δουλεύουμε χέρι με χέρι με την ε, υπατιαρμοστία αρμοστία προσφύγων του ΟΗΕ ε, και νομίζω ότι η συσχέτιση με τα Ηνωμένα Έθνη θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα να διεισδύσουμε στη Συρία. Τώρα, το άλλο θέμα ε, ε, είναι εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι και η σχέση με τους πολιτικούς γιατί πραγματικά ε, ίσως είναι και ευτυχές και όχι ατυχές το γεγονός ότι δεν μας προσέχουν ή δεν γνωρίζουν την πρωτοβουλία μας ε, γιατί ίσως αγνοούν την δύναμη που έχει η βιβλιοθήκη και τα βιβλία για να επηρεάσει τον κόσμο. Τώρα για τη λογοκρισία εμείς λέμε ότι οι εταίροι μας είναι αυτοί που θα επιλέξουν τα βιβλία και οι, και συνεργαζόμαστε για να γίνουν σωστές επιλογές. Δεν επιβάλλουμε κανένα βιβλίο. Θα φτιάξουμε ένα ηλεκτρονικό κατάλογο όπου αυτοί που θα συνεργαστούν μαζί μας θα μπορούν να διαλέγουν τίτλους αν θέλετε. Δύο πολύ πολύ σύντομες παρατηρήσεις να πω ότι η πρώτη βιβλιοθήκη χωρίς σύνορα φτιάχτηκε από τον πράγματι από τον ΕΣΕΛ και νομίζω ότι η μέθοδος και ο τρόπος εργασίας και λειτουργίας των βιβλιοθηκών χωρίς σύνορα ήταν να δουλεύουν σε τοπικό επίπεδο στενή συνεργασία με δημιουργούς και άλλους. Τώρα για αυτούς με τα προβλήματα όρασης. Στην Ασία ε, έγιναν, ε, έγινε υποδειγματική δουλειά από ομάδες ε, Γάλλων που πραγματικά βοήθησαν. Ε, μια κυβερνητική οργάνωση ήταν ε, αυτοί οι Γάλλοι, ε, έκαναν εξαιρετική δουλειά και μακάρι να γίνουν και να συνεχιστεί η δουλειά αυτή. Να πω και εγώ κάτι τι. Θα ξέρετε σίγουρα ότι το 2015 ε, φτάνουμε θα πρέπει να δούμε και τους στόχους της ε, χιλιετίας πραγματικά τι επετέφθη από αυτούς ε, κάπου ε, οι βιβλιοθήκες και η άτυπη εκπαίδευση ε, παραμελήθηκαν λίγο και ειλικρινά νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να καθίσουμε να ξανασκεφτούμε γιατί η άτυπη εκπαίδευση είναι σημαντική και εκεί μπορούν να βοηθήσουν ε, τα ευρωπαϊκά όργανα γιατί εδώ μιλάμε για πρόσβαση στη γνώση και νομίζω ότι πρέπει να υπήρχαν τέτοιοι στόχοι στα, στους στόχους χιλιετίας και για την περίοδο μετά το 2015 θα πρέπει να επαναληφθούν. Ναι. Να σας πω ότι οι βιβλιοθήκες χωρίς σύνορα λειτουργούν και ε, στην Γαλλία και εκτός ε, προφανώς ε, αλλά και στη Γαλλία λειτουργούμε παρόλο που ίσως δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Πρόεδρο, συγγνώμη, συγγνώμη που αναγκάζομαι να κόψω τη συζήτηση. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και ελπίζουμε να ε, έρθετε σε επαφή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχει σχετικά κονδύλια για να μπορέσετε να έχετε και κάποια χρηματική στήριξη. Πάτε να δείτε τον Επίτροπο Πίμπαλξ πραγματικά. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που κάνετε.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 Uh, I Να καλωσορίσω έναν από τους πιο διακεκριμένους ε, ηγέτης που είχαμε από την Αφρική και μάλιστα παγκόσμιο ηγέτη. Περιμένουμε και τον κύριο Μπρόκ να έρθει, αλλά έχει καθυστερήσει. Όχι, να νάτος. Καταφτάνει. As we were Mr. His Excellency η αυτού εξοχώτης, ο κύριος Μπέκη, είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους ανθρώπους ε, ε, πολιτική προσωπικότητα της Αφρικής και έχει κάνει πάρα πολλά. Ε, είναι γνωστά τα όσα έχει κάνει, μάχη κατά του Απαρτχάιτ, δύο θητείες ως πρόεδρος, βοήθησε την οικονομία της, Αφρική, της Νότιας Αφρικής, από το 4,5% το έπαινε και στο 6,5%. Είχε το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων επενδύσεων που ήρθαν στη διάρκεια της θητείας του στη χώρα και έκτοτε έχει κάνει και πάρα πολλές προσπάθειες σε ειρηνευτικές διαδικασίες σε άλλα τμήματα της Ιφρικής, συμπεριλαμβανομένου του Μπουρούντι, της ακτής του Ελεφαντοστού και βοήθησε φυσικά και στη μετάβαση της Αφρικανικής Ένωσης ε, σε αυτό που είναι σήμερα ένας πολύ ισχυρός οργανισμός ε, στην Αφρική, την ε, Αφρικανική Ένωση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα πλέον. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αλλάξει το ρούν της ιστορίας και έχει συνεισφέρει σημαντικά σε όλες τις ζω... στις ζωές όλες, όλων μας. Και είναι εδώ σήμερα για να συζητήσει μαζί μας κάτι εξίσου σημαντικό. Ε, στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτυσσόμενων χωρών έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το θέμα των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών από την Αφρική. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι είναι εδώ ως πρόεδρος του πάνελ υψηλού επίπεδου, της ομάδας υψηλού επίπεδου, γι' αυτό το τόσο ευαίσθητο ζήτημα και είναι ένα πολύ σημαντικό πρότυπο όχι μόνο για την Αφρική αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας από τους ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει στην επίσημη χρηματοοικονομική βοήθεια προς την Αφρική. Και επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω και τα μέλη της Επιτροπής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η πρόεδρος άλλωστε της Υποεπιτροπής είναι αυτή η οποία ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία ε, το περασμένο καλοκαίρι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι καλωσορίζω και τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Έλμαρ Μπροκ εδώ τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος ε, θα ε, συμπροεδρεύσει εδώ μαζί μου σε αυτή τη συνεδρίαση. Και θα ήθελα να δώσω λοιπόν τα ενία στον κύριο Μπροκ. Uh, κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπέκη, στο ίδιο, στην ίδια πλευρά του τραπεζιού όπως και εσείς ε, μετά τον Νέλσον Μαντέλα ε, για το θέμα των χρηματοοικονομικών ροών στην Αφρική ασχοληθήκατε ιδιαίτερα γι' αυτό επηρεάζει την οικονομική κοινωνική ανάπτυξη και τη δική σας και τη δική μας και ε, λέγεται ότι η, μιλάμε για ποσά το των 50 δις, δηλαδή διπλάσια κονδύλια α, σε σχέση με τα ποσά που παίρνει σε αναπτυξιακή βοήθεια η Αφρική. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται εδώ και πιο, πιο στενή και περισσότερη συνεργασία για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε κάπως τα πράγματα και τον Ιούνιο του 2013 οι ηγέτες του G8 αποφάσισαν ορισμένους κανόνες διαφάνειας που ισχύουν παγκοσμίω. Δεν είναι η Αφρική λοιπόν μοναχά στην οποία γίνονται παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Είναι ο κόσμος ολόκληρος. Εγώ πιστεύω όμως ότι ειδικά με τις αφρικανικές κυβερνήσεις πρέπει να ε, συνεργαστούμε περισσότερο για να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι σε σχέση με αυτές τις ροές. Έχετε το λόγο. Ε, ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους δύο συμπροέδρους και τα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα διότι μας δίνεται χρόνο να σας μιλήσουμε για αυτά τα οποία ανέφεραν οι συμπρόεδροι για ένα τόσο σημαντικό θέμα λοιπόν. Το θέμα των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών από την Αφρική. Η ομάδα μας ε, συστήθηκε ως αποτέλεσμα των ε, συμφωνιών των Υπουργών ε, Οικονομικής Ανάπτυξης στην Αφρική, οι οποίοι προσπάθησαν να κινητοποιήσουν εσωτερικούς πόρους στην Αφρική προκειμένου να βοηθήσουν τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Και ακριβώς αυτό το πλαίσιο προέκυψε και το ζήτημα αυτό. Η Αφρική έχανε σημαντικούς πόρους τους οποίους χρειάζεται προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει αυτή την ανάπτυξη. αν ε, ποσά δισεκατομμυρίων και αυτά τα ποσά ε, θεωρούνται και συντηρητική εκτίμηση των πραγματικών ε, ροών που φεύγουν από την Αφρική. Πρόκειται λοιπόν για πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό το οποίο ε, αναμένεται να κάνει η ομάδα μας είναι εν τέλει μέχρι τον Ιούνιο-Ιούλιο του τρέχοντος έτους να υποβάλει μια έκθεση ε, στην οποία θα κάνει συστάσεις προς τους επικεφαλείς μας που είναι οι υπουργοί οι οποίοι από εκεί και πέρα θα ε, αναφέρουν στην Σύνοδο της Αφρικανικής Ένωσης συστάσεις λοιπόν για το τι θα πρέπει να κάνει η Αφρική για το ζήτημα αυτό αλλά επίσης και συστάσεις για το τι θα πρέπει να κάνει ο υπόλοιπος κόσμος για το ζήτημα διότι ε, όπως γνωρίζουν όλοι, οι πόροι αυτοί φεύγουν παρανόμως από την Αφρική αλλά κάπου καταλήγουν. Επομένως υπάρχει μια χώρα παραλήπτης, ένας φορέας παραλήπτης, κάποιος κάπου τα παίρνει αυτά τα χρήματα. Επομένως είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε και τις δύο πτυχές του ζητήματος και αυτό σημαίνει ότι προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα χρειαζόμαστε και συνεχή συνεργασία. Γι' αυτό ακριβώ και ήταν σημαντικό να έρθουμε εμεί εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολείται με το ίδιο πρόβλημα και όπως αναφέρθηκε, ε, το θέμα αναφέρθηκε και στην τελευταία συνεδρίαση του G8, ε, όχι απλώς ως ένα θέμα το οποίο αφορά την Αφρική και τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά ως παγκόσμιο πρόβλημα. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι ως προς το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολούνται με τα θέματα αυτά, γι' αυτό και θεωρήσαμε ότι είναι απαραίτητο να έρθουμε εδώ και να σας συστηθούμε, διότι χρειαζόμαστε αυτή τη συνεργασία. Αν μου επιτρέπουν εδώ οι δύο προεδρεύοντες, θα ήθελα να ζητήσω από, τον συνάδελφο, από τη συνάδελφο να σας ε, κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Ευχαριστώ εξοχότατε και εκ μέρου των συναδέλφων μου να πω ότι αποτελεί τεράστια τιμή για εμάς που μας δίνετε το βήμα να ε, συζητήσουμε για το ζήτημα των παρανόμων ε, χρηματοοικονομικών ροών. Θα ήθελα επιγραμματικά να σας δώσω μια παρουσίαση της κατάστασης, το πάνελ, όπως είπε και η εξοχότητά του, ασχολείται με το ζήτημα αυτό πάνω από ένα χρόνο. Λάβαμε την εντολή να ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό με το, από το Συμβούλιο Υπουργών της Αφρικανικής Ένωσης και όπως είπε και ο κ. Μπάκη, αντιλήφθη το Συμβούλιο Υπουργών την σημασία του προβλήματος, καθώς επίσης και τη σύνδεση αυτού του προβλήματος με τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις της Αφρικής. Κατά βάση, οι παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, όπως εμείς τις ορίζουμε, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων στην Αφρική και δεδομένης της ε, γνώσης και του θέματα, των θεμάτων με τα οποία ασχολείται η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιλαμβάνεστε πολύ καλά τι εννοώ. Οι αριθμοί, οι εκτιμήσεις κυμαίνονται από 22 δισεκατομμύρια από το 2008 ε, το χρόνο αλλά φτάνουν μέχρι το 200, 2008 πλέον μιλάμε για πλέον κοντά στα 50 δισεκατομμύρια. Αυτού του είδους η αφέμαξη των οικονομιών έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο ΑΕΠ, στην χρήση, στην κατανομή των πόρων στην Αφρική. Πρόκειται λοιπόν για απώλεια πόρων, όχι απώλεια πόρων που ε, ε, δεν υφίσταντο, αλλά ουσιαστικά για κακή χρήση των πόρων που υπάρχουν. Αν μιλάμε για 50 δισεκατομμύρια. Και το διαρέσουμε με τον αριθμό των αφρικανικών χωρών. Πρόκειται για ένα δισεκατομμύριο το χρόνο για κάθε αφρικανική χώρα. Αυτό είναι τεράστιο, εάν λάβουμε υπόψη μας τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους για επενδύσεις στον τομέα της ανάπτυξης Η κυβερνησει Η εντολή που έχει δοθεί στο πάνελ είναι συγκεκριμένη. Θα πρέπει να ε, εξορίσει το, το, το, το επίπεδο, να ορίσει τι είναι οι χρημα, παράνομες χρηματοοικονομικές ροές, ποια μοτίβα ακολουθούνται, ποιο είναι το επίπεδο του, να εκτιμήσει ποιες είναι οι περίπλοκες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις αυτών των ροών, καθώς επίσης και να ευαισθητοποιήσει τις αφρικανικές κυβερνήσεις, καθώς επίσης και άλλους φορείς, που είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ, να ευαισθητοποιήσουμε τις κυβερνήσεις, τους πολίτες, αλλά και τους εταίρους μας στην αναπτυξιακή συνεργασία. Και τέλος, να προτείνουμε συγκεκριμένες ε, πολιτικές και να κινητοποιήσουμε ε, φορείς οι οποίοι θα υποστηρίξουν αυτήν την, τις συγκεκριμένες πολιτικές για την καταπολέμηση των παράνομων οικονομικών ροών. Ο ορισμός που δίνουμε εμείς στο πάνελ αναφέρεται σε ε, χρήματα τα οποία έχουν παρανόμως αποκτηθεί, μεταφερθεί ή χρησιμοποιούνται παρανόμως. Και ιδιαίτερα αυτό σε ένα διακρατικό πλαίσιο. Το πάνελ λοιπόν εξετάζει όλων αυτών των ειδών τα ζητήματα και ήδη έχουμε επικοινωνήσει με άλλους φορείς το τελευταίο ένα χρόνο σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο στην Αφρική δεν ε, καταφέραμε να επισκεφτούμε κάθε χώρα, αλλά είχαμε ένα αρκετά προσωπευτικό δείγμα που μας έδωσε μια καλή εικόνα του τρόπου με τον οποίο ε, εκφράζεται το πρόβλημα στις διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, εξετάσαμε την ε, κατάσταση σε χώρες οι οποίες βρίσκονται σε σύνοπλε συγκρούσεις, όπως για παράδειγμα η Λιβερία, ή σε χώρες στις οποίες η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι πολύ σημαντική, όπως για παράδειγμα η λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Είχαμε λοιπόν ένα δείγμα 4-5 ε, κρατών από την ε, Αφρική και ε, επικοινωνήσαμε όχι μόνο με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αλλά επίσης και με τα Υπουργικά Συμβούλια των Κυβερνήσεων αυτών των χωρών. Επίσης με μέλη και της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας ενώ ταυτόχρονα είχαμε επαφές και με μη κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, τράπεζες αλλά επίσης και την κοινωνία των πολιτών γιατί θεωρούμε ότι στο ζήτημα αυτό χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την ευαισθητοποίηση και ο ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων και τέτοιου τύπου φορέων είναι εξαιρετικά σημαντικό προκειμένου να υπάρξει αυτή η ευαισθητοποίηση, να υπάρξει μια διάδοση τη πληροφορία και να υπάρξει σχετική κινητοποίηση. Στο πλαίσιο των περιφερειακών ε, ε, διαβουλεύσεων, μέχρι στιγμή ε, αξιοποίησαμε τι εξωτερικέ διαβουλεύσει, γιατί όπως είπε και η ψυχότητά του, χρειαζόμαστε συνεργασία και θα χρειαστεί να αναλάβουν δράση οι κυβερνήσεις της Αφρικής, αλλά επίσης χρειάζεται η υποστήριξη και των κυβερνήσεων της Ευρώπης αλλά και αλλού. Καθώς επίσης και η δράση από διακυβερνητικούς, διεθνεί φορείς. Ε, συνομιλήσαμε λοιπόν με την Αμερικανική κυβέρνηση, με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς επίσης και με τον ΟΑΣΕ και ε, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό βρισκόμαστε και εδώ και σας ευχαριστούμε γι' αυτό όπως είπε και ο πρόεδρος Μπέκη, χρειάζεται να εξετάσουμε το ζήτημα από δύο πτυχές. Πρώτον, την πηγή, από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα, η πηγή αυτών των χρημάτων στα κράτη της Αφρικής, αλλά επίσης και πού κατευθύνονται, προς τα πού πηγαίνουν. Γνωρίζετε, φαντάζομαι, ότι υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο διάφορες οντότητες, διάφοροι φορείς, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο και διευκολύνουν αυτές τις παράνομες χρηματοοικονομικές ε, ε, ροέ. Φορολογική παράδειση σε διάφορα σημεία του κόσμου, εκεί καταλήγουν πολύ συχνά αυτά τα χρήματα. Και συχνά έχουμε το φαινόμενο μια εταιρεία να φαίνεται ως ε, καθόλου ανόμιμη και νομότυπη, αλλά στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται ως βιτρίνα για την εξυπηρέτηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών. Προτείνουμε λοιπόν μια σειρά δράσεων που θα μπορούσαν να αναλυφθούν και στην Αφρική και εκτός. Η έρευνα που έχει διεξαχθεί επί χρόνια στο θέμα αυτό και το πάνελ μας αξιοποιεί την ήδη αποκτηθή γνώση, είναι ότι υπάρχουν δύο συστατικά στοιχεία αυτών των ροών. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια, ένα σύνολο συναλλαγών που έχουν σχέση με τη διαφθορά. Δηλαδή ε, παράνομα αποκτηθέντα από ακλοπές ή απάτες ή ουσιαστικά ε, ε, ε, διαφθορά. Υπάρχει επίσης ένα σύνολο συναλλαγών που έχει σχέση με εκβιασμούς, με πλαστογραφίες, με τέτοιου τύπου απάτες, το οποίο ανέρχεται στο 35% του συνόλου και μια τρίτη ομάδα συναλλαγών που ίσως εκπλήξει όσους δεν έχουν σχετική γνώση του θέματος, αλλά είναι σημαντική. Ένα ε, μέρος των διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Για παράδειγμα, υπερτιμολογήσεις, πλαστά τιμολόγια με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης και με βάση τα δεδομένα αυτό το ο τρίτο πυλώνα, αυτό το τρίτο σύνολο συναλλαγών καλύπτει το 65% του συνόλου. Συνήθως σκεφτόμαστε ότι το σημαντικότερο στοιχείο θα ήταν η διαφθορά και ε, μίζες ουσιαστικά, διαφθορά κρατικών αξιωματούχων, αλλά δεν, τα στοιχεία μας δείχνουν ότι υπάρχει και το υπόλοιπο 65% που είναι εξίσου σημαντικό. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε όλα τα στοιχεία και όλους τους παράγοντες που διευκολύνουν αυτές τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που εξετάζει το πάνελ είναι ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο προφανώς ενδιαφέρει τους πολίτες και πιστεύω ότι γι' αυτό είναι και εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα να απευθυνθούμε σε κοινοβούλια όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί τα κοινοβούλια εκπροσωπούν τους πολίτες. Είναι λοιπόν σημαντικό να εκτιμήσουμε και να γνωρίζουμε ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος αυτών των ροών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Μπορεί να φαίνονται υπερβολικά τεχνικά αυτά τα θέματα και μπορεί να μην γίνονται απολύτω ε, κατανοητά. Αν κάποιο δεν έχει ειδικέ γνώσει στον τραπεζικό τομέα, στη λογιστική, σε οικονομικά θέματα, μπορεί να μην καταλάβει ακριβώ ε, ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά για να βρούμε λύσεις έχουμε αντιληφθεί ότι μιας και πρόκειται για ένα ζήτημα συστημικό, για ένα πρόβλημα που αφορά σε συμφέροντα ή στις, στη, στη διαπλοκή και στη σχέση των διαφόρων ομάδων συμφερόντων, πρόκειται για αυτόν τον λόγο και για ένα εξαιρετικά πολιτικό θέμα. Άρα χρειάζεται να αντιμετωπιστεί και στο πολιτικό επίπεδο και στο τεχνικό επίπεδο. Προσπαθούμε λοιπόν μέσω της εκθεσής μας να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα διευκολύνει, θα επιτρέπει σε κάποιον να καταλάβει και το την πολιτική διάστηση του προβλήματος, ποιος είναι ο αντίκτυπος για παράδειγμα αυτών των συναλλαγών, αλλά επίσης και το τεχνικό στοιχείο, με ποιον τρόπο ε, γίνονται αυτές οι συναλλαγές και ποιες δράσεις μπορεί να αναλυφθούν από τις κυβερνήσεις και από άτομα. Τέλος, κλείνοντας για να τονίσω για άλλη μια φορά την σημασία των παράνομων ροών. Αυτές οι παράνομες ροές συμβάλλουν ή μάλλον προκαλούν σε σημαντικό βαθμό το χαμηλό βιωτικό επίπεδο και την χαμηλή αριθμό ανάπτυξης που παρατηρούμε στην Αφρική. Πρόκειται για έναν από τους λόγους που οι κυβερνήσεις της Υπήρου δεν καταφέρνουν να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς στόχους που θέτουν. Όχι μόνο τους στόχους που τίθενται σε εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης και σε διεθνές επίπεδο, όπως για παράδειγμα τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας. Μειώνεται, για παράδειγμα, η δυνατότητα μιας χώρας παραγωγής ε, ακαθαριστού εγχώριου προϊόντος, παραγωγής πλούτου, και αυτό οδηγεί στο να μην υπάρχει αρκετή τόσο, ε, αρκετά χρήματα για επενδύσεις στην υγεία, στην εκπαίδευση, σε έργα υποδομής. Οδηγεί επίσης και σε μείωση των φορολογικών εσόδων. Και αυτό ίσως είναι και ένα, ε, ε, ένα επιχείρημα που δείχνει ότι αυτά τα φορολογικά έσοδα, αν υπήρχαν, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τις κυβερνήσεις για αναπτυξιακούς στόχους. Όταν λείπουν αυτά τα φορολογικά ε, έσοδα, ε, αναγκαστικά οι κυβερνήσει αυξάνουν τη φορολογία των πολιτών. Και αυτά τα έσοδα θα μπορούσαν να βοηθήσουν ένα κράτος να έχει περισσότερους πόρους στη διάθεσή του για την υλοποίηση των εθνικών του πολιτικών εξαιτία τη φύση των φορέων που συμμετέχουν σε παράνομε χρηματοοικονομικέ ροέ, αυτέ οι ροέ εντείνουν την φτώχεια και την ανισότητα. Η μεγαλύτερη ανισότητα ενισχύει την ανισότητα, γιατί οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Κάτι που περιορίζει και τις δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα να αναπτυχθεί σε μια χώρα, σε εθνικό επίπεδο όπως είπα, υπονομεύει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, που μετά έχουν με τη σειρά τους ε, αυτά τα προβλήματα, άλλες επιπτώσεις. Και επίσης εξαιτία της φύσης αυτών των συναλλαγών διευκολύνεται η διαφθορά. Και η διαφθορά είναι ένα θέμα που πρέπει να μετωπιστεί και από την πλευρά την κρατική, δηλαδή των κρατικών αξιωματούχων, αλλά και των εταιριών ή οποιοδήποτε άλλων φορέων εμπλέκονται σε εθνικό ή διεθνές ε, ή πολυεθνικό πλέον επίπεδο. Αυτέ οι παράνομε ροέ επίση έχουν συμβάλει στην αύξηση του εξωτερικού χρέου τη Αφρική. Κάτι που υπονομεύει την δυνατότητα των κρατών. Και αυτή η Διαφθορά υπονομεύει επίση και το κράτο δικαίου, τη δυνατότητα δίωξη των ενόχων, τη δυνατότητα λειτουργία του δικαστικού συστήματο, το κράτο δικαίου σε μια χώρα γενικά. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που μας δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσουμε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του εξαιρετικά σημαντικό αυτό ζήτημα. Θεωρούμε ότι σε συνεργασία με φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με τρόπο αποτελεσματικό, γιατί ως Κοινοβούλιο έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην νομοθεσία και στην λογοδοσία και μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτόν τον ρόλο έτσι ώστε να ενισχυθεί και το κανονιστικό πλαίσιο και να ε, η λογοδοσία. Για παράδειγμα, ένα κανονιστικό πλαίσιο για τις διεθνείς συναλλαγές, για τις διακρατικές συναλλαγές, για τον τραπεζικό τομέα, που να ενισχύει την διαφάνεια, έτσι ώστε τελικά να προστατεύεται το συμφέρον του απλού πολίτη και στην Αφρική και στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Uh, we should give the floor to Mrs. Lochbieler. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Λόχ Μπίλερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε και για την παρουσίαση αυτή. Πραγματικά, αν μπορούσαν όλοι αυτοί οι πόροι να παραμείνουν στην Αφρική, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ε, σωστές επενδύσεις στην παιδεία, στην... Ε, ε, υγεία λοιπά. Εγώ προέρχομαι από την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ε, θα με ε, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με την εξορυκτική βιομηχανία, παραδείγματο χάρη στην Αγγόλα. Έχω λοιπόν μια ερώτηση για το έκθεση που ετοιμάζεται. Θα ζητήσετε να ενισχυθούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιμένουν να υπάρχει λογοδοσία και διαφάνεια στον τομέα παραδείγματος χάρη εξοριστικής βιομηχανίας πρώτων υλών ή το παράδειγμα της Αγκόλας μας έδειξε πόσο δύσκολο είναι να διεισδύσουμε στον τομέα αυτό. Ρόμπερτ Άκκινς. Ευχαριστώ πρόεδρε ή πρόεδροι στον πληθυντικό θα έπρεπε να πω με εγωιτεύει το θέμα διότι δεν ήξερα πολλά πράγματα έχω λοιπόν αρκετές ερωτήσεις αυτό το αυτά τα χρηματικά ποσά είναι πολύ μεγάλα φαντάζομαι ότι καταλήγουν σε κάποια τράπεζα δεν μπορούν να ανακαλυφθούν. Άμα χάσει κανείς 500 ευρώ μπορεί να μην το πάρει κανείς είδηση αλλά 50 δις είναι τεράστια ποσά για τα οποία κάποιος κάτι πρέπει να ξέρει και θα πρέπει να μπορούμε να τα βρούμε αυτά κονδύλια τι είναι επίσης, είναι μετρητά, είναι χρυσός, είναι ομόλογα, τι είναι, είναι άνθρωποι με βαλιτσούλες γεμάτες χρήματα που κυκλοφορούν και τα 50 δις τι είναι, είναι πολλές συναλλαγές ε, που κάποιες, λίγες μεγάλες συναλλαγές όμως που γίνονται μέσω διαδικτύου είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρουν τα βαλιτσάκια και τι εξουσία έχουμε σε, έχετε μάλλον σε σχέση με τις κυβερνήσεις κάποιων αφρικανικών χωρών ε, ούτως ώστε να μπορείτε να κάνετε κάτι. Συγγνώμη που θέτω όλα αυτά τα ερωτήματα δεν νομίζω ότι ε, και συγγνώμη που έχω τόσες ερωτήσεις κανείς δεν μου πρόσφερε και τίποτα από όλα αυτά τα ποσά θα ήθελα όμως να ξέρω και πραγματικά με, ε, θα ήθελα να μάθω λεπτομέρειες και να μου πείτε και τι μπορείτε εσείς να κάνετε για αυτά Thank you, Mr. Um, Ευχαριστώ πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια οδηγία διαφάνεια για την εξορρυκτική βιομηχανία όπου προσπαθούμε να επιβάλλουμε εκεί περισσότερη διαφάνεια από ό,τι υπήρχε στο παρελθόν με μια έννοια αντιγράφουμε το νόμο των Φρανκ των Αμερικανών λοιπόν πιστεύετε εσείς ότι οι νομοθετικές μας πρωτοβουλίες κάνουν αρκετά μήπως πρέπει να πάμε λίγο παραπέρα. Αυτή είναι η στιγμή για να μας πείτε τι, τι νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω από νομοθετική άποψη για να βοηθήσουμε στο θέμα αυτό. <laughs> Η κυρία Γκόμες σήμερα έχει και γενέθλια, 45 χρονών γίνεται. Συν 15 λέει η κυρία Γκόμες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που κάνατε και το ότι ακριβώς θέσατε το θέμα αυτό υπόψη μας για το οποίο πρέπει να συνεργαστούμε. Πρέπει να συνεργαστούμε βέβαια σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά αν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αφρικανική Ένωση ήδη κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Η κυρία Λόχφιλερ τόνισε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο κάναμε μια έκθεση για το πώς μπορούμε να μετρήσουμε τη διαφθορά σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και πραγματικά εκεί έχετε πάρα πολλά προβλήματα οφείλω να πω αλλά χρειάζεται βέβαια και στήριξη και συνεργασία. Ε, το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή ασχολείται με την αναθεώρηση της οδηγίας για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό αυτό και θα ζητήσουμε ε, πολλά πράγματα στην καινούργια αυτή ε, οδηγία. Πολλά πράγματα μπορούν να βοηθήσουν και εσάς. Τα μέλη της Αφρικανικής Ένωσης τι κάνουν. Α, να σας πω, οργανώθηκε την περασμένη εβδομάδα μια... Ε, τη δημόσια ακρόαση με έναν δημοσιογράφο που ήρθε από την Αγγόλα και που και μία κυρία που της οποίας οι δύο γη σκοτώθηκαν στην Αγγόλα δεν μπορούσε να κάνει τίποτε στη χώρα της ήρθε στην α, Πορτογαλία γιατί ήθελε πραγματικά να κάνει μια δημόσια καταγγελία και η συνάντηση του κυρίου Μπαρόζο, την κυρία Άστον κτλ. Τώρα η Πορτογαλία θεωρείται πλυντήριο για βρώμικο χρήμα και εκεί πραγματικά αγοράζεται και σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης ιδιαίτερα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Μια άλλη περίπτωση υπόθεση που συζητείτε αυτή τη στιγμή είναι η σημερινή Γουινέα που είναι άκρος διεφθαρμένη ε, και εγκληματική η ηγεσία της πρόσφεραν να αγοράσουν μία πορτογαλική τράπεζα η οποία διασώζεται αυτή τη στιγμή με ευρωπαϊκά κονδύλια ε. λοιπόν να αγοράσουν την τράπεζα αυτή γιατί για να έχουν ένα πλυντήριο, ένα τόπο να ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα τους. ερώτηση λοιπόν εσείς στην ομάδα υψηλού επίπεδου τι προτείνετε συγκεκριμένα στα μέλη της Αφρικανικής Ένωσης να κάνουν για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. vielen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται νομίζω να τονίσω και πάλι πόσο σκανδαλώδης είναι η κατάσταση που οδηγούν στη διαρροή, διαφυγή από την Αφρικανική Υπηρώ 50 δισεκατομμυρίων το, η Ευρώπη και τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τι μερίδιο έχουν σε αυτά τα χρήματα όπως είπαν και οι συνάδελφοι φεύγουν αυτά τα 50 δισεκατομμύρια αλλά καταλήγουν κάπου, κάπου πάνε και νομίζω ότι ξέρουμε όλοι που πάνε, σε ποιες χώρες, σε ποια ακίνητα επενδύονται και τα λοιπά. Ρωτώ λοιπόν γιατί δεν γίνεται τίποτε αυτή την ερώτηση πρέπει να τη θέσουμε βέβαια στους εαυτούς μας, ε. είναι ίσως λίγο αφελής. Από την άλλη μεριά είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρήματα αυτά, τα οποία παρήχθησαν παράνομα και διαφεύγουν από την Αφρικανική Ήπειρο παράνομα. Ρωτώ λοιπόν εσάς, τι θέλετε εσείς να κάνουμε για να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά στους ιδιοκτήτες τους. Ένα ερώτημα αυτό. Δεύτερο ερώτημα. Πω, κατά την άποψή σας, τι ποσοστό ή σε απόλυτες τιμές ε, τι πάνε στις σε ευρωπαϊκές τσέπες από αυτά τα χρήματα δεν ξέρω, μπορεί να είναι και μέσω εμπορικών ροών, να υπολογίζονται λάθος κάποιες τιμές ή μπορείτε να μας δώσετε μερικές λεπτομέρειες. Και επανέρχομαι στο ερώτημα, πείτε μας τι θέλετε να κάνουμε. Θέλετε νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ή απλώς αρκεί να εφαρμόσουμε καλύτερα τις υφιστάμενες νομοθετικές πράξεις. Κατά την άποψή σας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς εδώ. Ε, εμείς σαν ε, ευρωβουλευτές. Ε, κυρία Τεκέζερ, συγγνώμη δεν άκουσα που φωνάζετε το όνομά μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε Μπέκη, για τις ομάδες υψηλού επίπεδου επιλέγετε πάντα δύσκολα ζητήματα. Εγώ σας είχα γνωρίσει στη συζήτηση για τον Νότιο Σιουδάν και τώρα βρίσκεστε επικεφαλής ένα ως προβλήματος που είναι τουλάχιστον εξίσου περίπλοκο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Πραγματικά χρειαζόμαστε όλοι πολύ τύχη. θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από πλευράς Αφρικανικής Ένωσης ε, και είναι δίκαιο το γεγονός ότι συστήθηκε μια ομάδα υψηλού επίπεδου που προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα. Και νομίζω ότι ε, ενδιαφέρει σίγουρα και αφρικανικές ε, κυβερνήσεις και ευαισθησίες, αλλά όπως ακούστηκε και πολυεθνικές και μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αλλά και ευρωπαϊκά κράτη. Δεν μπορεί τα πράγματα να είναι άσπρα από τη μία και μαύρα από την άλλη. Επιτρέψτε μου αυτό το λογοπαίγνιο, τουλάχιστον από πλευράς ε, δεοντολογίας και και μόνον. Ε, νομίζω ότι αν τα ψάξουμε θα είναι δύσκολα τα πράγματα κατέρωθεν. Και φυσικά σίγουρα θα σας υποστηρίξουμε από αυτού και δεν ε, θα σας ζητήσουμε περισσότερα από όσα μπορείτε να μας δώσετε σήμερα, γιατί μόλις ξεκινάει η συζήτηση για το θέμα. Αλλά θα ήθελα να σταθώ λίγο στο θέμα του Νοτιού Σιδάν, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά, διότι πρόκειται για μια πολύ νέα χώρα, μόλις δημιουργήθηκε και ευθύς εξ αρχής φαίνεται ότι ε, είχε πολύ σημαντικές περιπτώσεις διαφθοράς ε, για τις οποίες ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε ουσιαστική βοήθεια και θα ήθελα, ίσως επειδή γνωρίζετε το ζήτημα, να μας πείτε λίγο τι έλειψε από πλευράς ευρωπαϊκής. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη δημιουργία αυτού του κράτους, Στην οικοδέματα ενός ε, νέου κράτους ε, και τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε. Όταν είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλά χρόνια ζωής, φυσικά δημιουργεί τη διαφθορά, είναι κάτι το οποίο είναι δρεωμένο, είναι περίπλοκα τα πράγματα, αλλά εδώ ζητούμε περισσότερη διαφάνεια, μπορούμε να έχουμε περισσότερο έλεγχο. Τι άποψη έχετε εσείς για αυτή την περίπτωση, την τόσο συγκεκριμένη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας. Ο κύριος Ντέβα. Επιτρέψτε μου και εμένα να σας θέσω μια ερώτηση. Υπάρχει αυτή η έκφραση ότι χρειάζονται δύο για να χορέψουν ένα ταγκό. Δηλαδή τα πάντα είναι θέμα συνεργασίας. Ε, δεν μπορεί να βρεθούν ξαφνικά βαλίτσες με χρήματα στο κρεβάτι κάποιου στην Ευρώπη. Κάποιος τα έφερε. Υπήρχε μια υπόθεση όταν εγώ έμεινα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο και ήθελαν να βρούνε που βρίσκονται τα χρήματα του Πρόεδρου Αμπούντα. Και τα βρήκαμε. Ήτανε... Και ήταν στη Βικτόρια στην τράπεζα Barclays. Και φυσικά ήταν πολύ δύσκολο το θέμα γιατί ο Διοικητικό Συμβούλιο της Barclays, αλλά τελικώς τα χρήματα ήταν σε μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Κάπου πρέπει να είναι λοιπόν αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να είναι κρυμμένα κάτω από το μαξιλάρι του καθενός. Και τι γίνεται λοιπόν με τον άλλο, ε, τον ε, ε, συνοδό στο ταγκό. Και τι γίνεται με τις τράπεζες, πώς συνομιλείτε με τις τράπεζες, τις τράπεζες του Λιχτενστάιν, της Ελβετίας ή του Λουξεμβούρου. Θα μπορούσα να συνεχίσω τον κατάλογο, αλλά έχουμε πολλές τράπεζες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ναι. Well, I... Η κυρία Σαρχεντίνη. Νομίζω ότι εγώ με κάποιες από τις ερωτήσεις που ετέθησαν και κάποιες παρατηρήσεις του κυρίου Στέρντι και του κυρίου Ντέβα θα μπορούσα ίσως να συνεχίσω ως εισηγήτρια της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών για την τέταρτη αναθεώρηση της νομοθεσίας για την νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων. Είχα την τιμή να συζητήσω με τον πρόεδρο Μπέκη και την Επιτροπή του νωρίτερα σήμερα και Ε, από τις εξηγήσει που δόθηκαν, που νομίζω ότι καλό θα ήταν να ακούσετε και εσείς εδώ, φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη πλειοψηφία που είναι υπέρ ενός ε, μητρώου για τους τελικούς δικαιούχους. Ε, θα ψηφίσουμε μάλλον την επόμενη εβδομάδα, αλλά φαίνεται ότι όλο το φάσμα των πολιτικών ομάδων συμφωνεί για ένα δημόσιο μητρό και στα 28 κράτη-μέλη, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο διαδικτυακά με ανοιχτά δεδομένα δημόσια σε όλους δεν θα υπάρχει κανένας περιορισμός. Και για μένα αυτό προσωπικά ε, είναι πολύ καλά νέα, όχι μόνο για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης εγκληματικών δραστηριοτήτων, αλλά ε, προκειμένου και η κοινωνία των πολιτών ε, επιτρέψτε μου την έκφραση, να ξεκαθαρίσει λίγο την κοινωνία της για τις έρευνες των δημοσιογράφων, να μπορούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις να βρίσκουν ε, τις ε, ε, ε, κρυμμένες επιχειρήσεις, τις ε, επιχειρήσεις που κρύβονται πίσω από άλλη επωνυμία, ε, η μία πίσω από την άλλη και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διοχετεύουν χρήματα. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο εσωτερικό μας ζήτημα, είναι παγκόσμιο, αλλά αν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 28 κράτη-μέλη δώσουν ε, ένα παράδειγμα και υπάρχει ένα μητρό τελικών δικαιούχων, θα δώσουν ίσως και ε, ένα καλό παράδειγμα για τους υπολείπους. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι θα ήταν καλό να συνειδητοποιήσουμε εμείς εδώ στην αίθουσα, αλλά φυσικά και η ομάδα του Προέδρου Μπέκη είναι ότι αυτό φυσικά είναι μόνο το ίμιση της νομοθεσίας. Χρειαζόμαστε και τα κράτη-μέλη στο πλευρό μας. Έχουμε τον Πρόεδρο του Καμερού, ε, τον... Ε, συγγνώμη, τον πρόεδρό σας, τον κύριο Κάμερον, κύριε Ντέβα, αλλά φαίνεται ότι οι Γερμανοί ε, εξετάζουν ακόμα το ενδεχόμενο της δυνατότητας να υπάρχει αυτό το δημόσιο μητρό. για να μπορέσουμε να καταπονομήσουμε τις παράνομες χρηματοοικονομικές ε, ροές από την Αφρική θα πρέπει τουλάχιστον εμείς να ξεκαθαρίσουμε τα εσωτερικά μας ζητήματα και να μην είμαστε ασφαλείς λιμένας ε, για κονδύλια τα οποία χάνονται και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις σε υποδομές, σε σχολεία, σε δρόμους στην Αφρική. Και όχι μόνο λοιπόν να προσφέρουμε ηθική υποστήριξη στην ομάδα υψηλοπιπέδου του Πρόεδρου Μπέκη, αλλά θα μπορούσαν οι συνάδελφοι να προσπαθήσουν να επηρεάσουν και τις ίδιες τους τις κυβερνήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αν κατάλαβα καλά, αυτό που λέμε είναι ότι θα υπάρξει ένα μητρό στο οποίο θα καταγράφονται όλε οι συναλλαγέ στην Ευρώπη. η κυρία Αργεντίνη. Θα, ονειρευμένο θα ήταν αυτό, αλλά δεν ζητάμε κάτι τέτοιο. Στο πλαίσιο τη ε, νομοθεσία για την καταπολέμηση του ξεπλήματο μαύρου χρήματο, καθώ επίση και την καταπολέμηση τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, οι ε, διάφορες οντότητες όπως για παράδειγμα οι τράπεζες ή ένα καζίνο ή κάποια ε, ε, real estate κάποιος που κάνει επενδύσεις σε ακίνητα θα είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει ποια είναι η προέλευση των χρημάτων που επενδύθηκαν ή δόθηκαν σε αυτούς. Και μετά αυτό το μητρό θα είναι υποχρεωμένα ναι, αυτές, οι, αυτές, αυτοί οι να τον συμπληρώνουν και θα είναι διαθέσιμο, δημοσιοποιημένο και προσβάσιμο και στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό λέμε. Ο κύριο Μποκ και ποια είναι η κοινωνία των πολιτών, απάντησε τη κυρία Σαρτζετίνη, ε, εσείς και εγώ. Κύριος Μποκ, εγώ είμαι πολίτης, δεν είμαι κοινωνία των πολιτών. Κυρία Σαρτζετίνη, καλά, μπορούμε να την κάνουμε κάποια στιγμή αυτή τη συζήτηση. Αλλά ως εισηγήτρια χαίρομαι για το σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει σε αυτό το διάλογο. Εκτός μικροφώνου. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ζητήσω από τη συνάδελφο, την, ε, τον συνάδελφο κύριο Μπέικλορ να απαντήσει σε ορισμένες από τις ερωτήσεις. Ρωτάτε πώς γίνεται αυτή η μεταφορά των χρημάτων. Φεύγει από την Ήπειρο με βαλίτσες, ε, περπατάει, κολυμπάει, φεύγει με αεροπλάνα. Πώς πάει, πώς γίνεται όλο αυτό, με αυτά με ρωτάτε. Ήταν στοιχείο σε πολλές από τις ερωτήσεις των βουλευτών. Και μετά τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλα αυτά. Αλλά πρώτα θα ήθελα να εξετάσω κάποια άλλα ερωτήματα. Όταν η συνάδελφος ε, παρουσίασε την ε, μελέτη που έχουμε κάνει σε σχέση με την Αφρικανική Υπηρώ, είπε ότι σκοπεύουμε να εστιάσουμε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή τη συνεργασία με την ε, κοινωνία των πολιτών. Όποιο και αν είναι η κοινωνία των πολιτών, κύριε Μπόρκ. Θέλουμε να εμπλέξουμε την κοινωνία των πολιτών σε κάθε επίπεδο. Ε, στην βόρεια, ανατολική, δυτική, νότια, κεντρική Αφρική, παντού. Προσπαθούμε να τους ευαισθητοποιήσουμε, να καταλάβουν ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή θα κάνουμε τις προτάσεις μας, θα προτείνουμε συγκεκριμένες δράσεις. Μετά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει πίεση από κάτω. Να υπάρχει μια πίεση από τους πολίτες που θα αναγκάσει τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση. Και εκεί είναι που χρειάζεται η παρέμβαση της, πολιτείας, της ε, κοινωνίας των πολιτών. Γι' αυτό τον σκοπό έχουμε εντάξει στις δραστηριότητές μας την διαβούλευση και τη συζήτηση με την κοινωνία των πολιτών. Το θεωρούμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της δουλειάς του πάνελ. Ήταν από τις πρώτες μας πρωτοβουλίες να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, να τον ευαισθητοποιήσουμε και να συλλέξουμε οποιαδήποτε πληροφορία, η έκθεση, η στοιχεία, τα οποία θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ε, στην σύνταξη και της έκθεσης του πάνελ αλλά και στην προετοιμασία μας για το μέλλον, για τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα δράσης που τελικά θα συμφωνηθεί. Αυτά όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών. Τώρα επίσης ρωτήσατε ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ε, και της δράσης που θα αναλάβουν τα Αφρικανικά κράτη και η Αφρικανική Ένωση κτλ. Όπως σας είπα, η Επιτροπή μας δημιουργήθηκε και έλαβε την εντολή της από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης των Αφρικανικών των κρατών, των κρατών μελών της Αφρικανικής Ένωσης. Επομένως, εμείς πρέπει να αναφερθούμε, να παραδώσουμε την πρότασή μας σε αυτό το Συμβούλιο Υπουργών. Το τι θα γίνει μετά και μάλιστα δεδομένου ότι όπως είπε και ο, ο πρόεδρος χρειάζονται δύο για να χορέψει κανείς ταγκό, τι θα γίνει ως προς τον στο άλλο εταίρο σε αυτό το, μάλλον χορευτή σε αυτό το δαγκό. Όπως σας είπαμε, επισκεφτήκαμε μια σειρά αφρικανικών κρατών και επιλέξαμε ορισμένα κράτη για να γίνει μια μελέτη περίπτωση. Να εξετάσουμε συγκεκριμένα τι συμβαίνει, για παράδειγμα, στην Ιγυρία. Μάθαμε ορισμένα πράγματα από την Ιγυρία. Σκεφτήκαμε τη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό, πρόκειται να επισκεφτούμε την Αλγερία, τη Μουζαμβίκη το... και άλλες χώρες. Εκκρεμεί ακόμα μια επίσκεψη στον Μαυρίκιο και την Νότια Αφρική. Και προσπαθούμε να καταγράψουμε την κατάσταση ακριβώ στις χώρες αυτές όσον αφορά τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές Αφενό αλλά αφετέρου να δούμε και τι δράση έχουν αναλάβει οι κυβερνήσεις αυτών των κρατών, εάν έχουν αναλάβει κάποια δράση. Να δούμε ποια είναι η νομοθεσία αυτών των κρατών. Να δούμε τι είδου θεσμικά όργανα και κυβερνητικά όργανα υφίστανται και τι κάνουν και πόσο αποτελεσματικά είναι. Τι γίνεται επίσης από την πλευρά της αστυνομίας, της εισαγγελίας, των διοκτικών αρχών πώς διώκονται όσοι διαπράττουν τέτοιου τύπου αδικήματα. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτών των επισκέψεων τίθεται και το ζήτημα των συνεργασιών, των διακρατικών συνεργασιών, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι συχνά υπάρχει έλλειμμα συνεργασία. Μπορεί να υπάρχει ένα τμήμα τη κυβέρνηση, ένα τμήμα τη διοίκηση, το οποίο να γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση, αλλά να μην συνεργάζεται με το διπλανό του και ακόμα και αν υπάρχει νομοθεσία, εξαιτία αυτή τη ε, έλλειψη συνεργασία και επικοινωνία να μην μπορεί να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε μια χώρα και δεν θα πω το όνομα που θα μας πούν ότι δεν γνωρίζουμε ούτε καν πόσο χαλκό ε, εξάγουμε. Βασιζόμαστε στις εκθέσεις, στα στοιχεία που μας δίνουν οι μεταλλευτικές εταιρείες, οι εξορυκτικές εταιρείες οι οποίες φυσικά μπορούν να παραποιήσουν τα στοιχεία και να πούν ότι θέλουν. Ή μπορεί να επισκεφτούμε μια χώρα και να μας πούνε ότι εκδίδουμε αλλιευτικές άδειε, αλλά δεν γνωρίζουμε πόσο είναι τελικά η ποσότητα των ψαριών που αλλιεύονται στα εθνικά μας ύδατα, ούτε καν ε, για σκοπούς φορολόγησης ή ε, ε, συλλογής φόρων. Δηλαδή, μια αλληλευτική εταιρεία σε αυτή τη χώρα μπορεί να ισχυριστεί σήμερα δεν υπήρξε καθόλου ψαριά και απλώ θα του πιστέψουμε. Προσπαθούμε λοιπόν να χαρτογραφήσουμε την κατάσταση, να δούμε πώ ακριβώ λειτουργεί αυτό το φαινόμενο και όλα τα υπόλοιπα που σα ανέφερα. Και ελπίζουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα θα, δούμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαχείριση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων στην Ιγυρία. Ο τομέας των πετρελαιοπηγών στην Ιγυρία. Φυσικά βέβαια δεν μπορούμε να επισκεφτούμε και τις 54 χώρες. Γι' αυτό έχουμε επιλέξει ορισμένες. Έτσι ώστε στο τέλος, συμπερασματικά, να μπορέσουμε να πούμε στα κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης, στην Αφρικανική Ήπειρο, ότι αυτά τα βήματα προτείνει το πάνελ μας να ακολουθήσουμε, να κάνουμε όπως είπαμε ήδη, τελικά το θέμα θα παρεμπιευθεί στην ε, Γενική Συνέλευση ε, Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Αφρικανικής Ένωσης, στο Συμβούλιο, και εκεί θα ληφθούν οι αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή ληφθούν οι αποφάσεις, θα πρόκειται για πολιτική επίσημη της Αφρικανικής Ένωσης. Και από εκεί και πέρα αποτελεί αρμοδιότητα της Αφρικανικής Ένωσης να δημιουργήσει τους μηχανισμούς που θα την υλοποιήσει. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος της Επιτροπής. Ο ρόλος της Επιτροπής πρέπει να καταλήξει σε συστάσεις, τις οποίες θα παραδώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο που του της έδωσε την εντολή να το κάνει. Έτσι ώστε τελικά να πούμε ρητά στους, στους υπουργούς, στους αρμόδιους, ότι έτσι έχουν τα πράγματα, υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί και αυτό προτείνουμε. Και τώρα έχουμε στο ζήτημα του τι περιμένουμε, τι αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε σχέση, για παράδειγμα, για με αυτό που αναφέρατε για ένα δημόσιο μητρό των δικαιούχων είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Ότι στι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, υπάρχει νομοθεσία. Ε, είμαι σίγουρος ότι θα τα συζητήσουμε πιο διεξοδικά αυτά σύντομα. Τώρα με ρωτήσετε για τον Νότιο Σουδάν. πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε για τον Νότιο Σουδάν, προφανώς, είναι ότι κατά βάση και πρωτερχικά την ευθύνη για το μέλλον του κράτους αυτού την έχει η ηγεσία του. Είμαι βέβαιος ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωρίζουν την κατάσταση της ένοπλης σύγκρουσης στο Νότιο Σουδάν και το γεγονό ότι προήλθε από μια σύγκρουση ε, μεταξύ ομάδων στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος. Το οποίο δεν προήλθε από κάποιο είδους ε, συγκρούσεις στην κοινωνία μεταξύ δύο ομάδων κοινωνικών ή τίποτα τέτοιο. Πρόκειται απλώς για δύο φράξεις εντός του κυβερνώντος κόμματος που συγκρούνται μεταξύ τους. Και το λέω αυτό γιατί είναι μέρος της απάντησης στην ερώτημα που μου θέσατε και κάτι που είναι θεμελιώδης, πολύ βασική πρόκληση. Βεβαίω πρωταρχικά η ευθύνη βαρύνει εκείνους. Αλλά βεβαίω υπάρχει και μια ευθύνη για εκείνους τους φορείς ε, που δίνουν βοήθεια σε χώρες όπως το Σουδάν, όπως για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να απευθυνθεί ευθέω στην ηγεσία του Νοτιού Σουδάν και να πούνε ωραία, τώρα υπάρχει ένα ανεξάρτητο κράτος, τι πρόκειται να κάνετε. Πώς σκοπεύετε να κυβερνήσετε αυτό το νέο ανεξάρτητο κράτος, γιατί στην πραγματικότητα αυτή η σύγκρουση που δημιουργήθηκε στο επίπεδο της ηγεσία τώρα μας οδηγεί σιγά σιγά σε φίλιο πόλεμο, ενώ στην πραγματικότητα το ζήτημα είναι το μέλλον του Νοτιού Σουδάν. Και μια σύγκρουση μεταξύ εκείνων που θέλουν να ηγηθούν. για να βελτιωθεί η κατάσταση στη χώρα. Επομένω λέω ότι ίσως θα έπρεπε να ε, μας είχε απασχολήσει αυτό από την αρχή. Γιατί χωρίς μια τέτοια συζήτηση, χωρίς τελικά να υπάρχει μια ηγεσία σε μια χώρα μια κυβέρνηση σε μια χώρα η οποία να έχει ένα θετικό όραμα και να καταλαβαίνει τι χρειάζεται να γίνει και να μπορεί να το υλοποιήσει, πιστεύω ότι χωρί αυτό, χωρί μια τέτοιου τύπου κυβέρνηση, οποιαδήποτε άλλη επέμβαση, οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση μάλλον, δεν μπορεί να βοηθήσει. Στο πλαίσιο της ε, προσπάθειας ε, ειρήνευσης, έτσι ώστε να γίνει μια πολιτική διαδικασία στην οποία θα εμπλακούν όλα τα πολιτικά κόμματα, η κοινωνία των πολιτών, οι θρησκευτικοί ηγέτες, οι παραδοσιακοί ηγέτες, να γίνει μια διάσκεψη ώστε να συζητηθεί το μέλλον του Νοτιού Σουδάν. Θα πρέπει να συζητηθούν τα προβλήματα, τα ζητήματα που οδήγησαν στη, στο ξέσπασμα αυτού του εμφυλίου πολέμου. Αλλά είναι επίσης σημαντικό Όταν πια ξεκινήσει αυτή η διαδικασία διαβούλευσης, κάτι θα πρέπει να γίνει και για το κυβερνόν κόμμα. Πριν ξεκινήσουμε να συζητάμε. Γιατί διαφορετικά η διχόνοια και η διάσπαση του ιδίου του κυβερνώντος κόμματος θα μεταφερθεί στην ε, ειρηνευτική διαδικασία, στη διαδικασία των συνομιλιών και θα την οδηγήσει σε αποτυχία. Δηλαδή αυτό που λέω είναι ότι στο, το τι συμβαίνει στο κυβερνόν κόμμα στο Νότιο Σουδάν αντικατοπτρίζεται και επηρεάζει όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και της χώρας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το θέμα πρέπει όλοι να το θέσουμε στην, ε, στους ηγέτες του Νοτίου Σουδάν να συμφωνήσουμε τελικά δηλαδή προς τα πού θέλει να πάει το Νότιο Σουδάν και επίση προς τα πού πηγαίνει και το ίδιο αυτό το κυβερνών κόμμα ω πολιτικό οργανισμό. Γιατί το, το κίνημα απελευθέρωσης του Σουδάν στην πραγματικότητα βασίστηκε στον στρατό απελευθέρωσης του Σουδάν. Πράγμα που έχει οδηγήσει σε στρατιωτικοποίηση του πολιτικού κόμματος που σήμερα κυβερνά. Και ξαφνικά βρίσκεται με έναν εξάρτητο κράτο αυτό το κόμμα και πρέπει να ασχοληθεί με την ανάπτυξη, με τη δημιουργία εκπαιδευτικού συστήματο, σχολείων κτλ. Είναι πολιτικό κόμμα, αλλά έχει στρατιωτική δομή. Και αυτό επηρεάζει προφανώς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και το, την ποιότητα της διακυβέρνησης που μπορεί να ασκήσει. Τέτοιου τύπου ζητήματα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να βοηθήσουμε χώρες όπως το Νότιο Σουδάν. Ιδίως εμείς που ερχόμαστε απ' έξω για να βοηθήσουμε τον Νότιο Σουδάν να φτάσει εκεί που πραγματικά πρέπει. Ευχαριστώ. Ακούστηκε ένας αριθμός, 50 δις το χρόνο εξαφανίζεται από την Αφρική. Και τονίζω ότι αυτό είναι και τελείως συντηρητική εκτίμηση. Από εκεί και πέρα πρόκειται Εδώ όμως το νούμερο αυτό ξεχνάει το λαθρεμπόριο κάποιες εμπορικές συναλλαγές και λοιπά ε, παράνομες ή Δεν είναι λοιπόν, είναι συντηρητική εκτίμηση αυτό. Το πραγματικό νούμερο είναι πολύ πιο ψηλά. Ερώτηση τώρα, πού πάει ναι, τα χρήματα αυτά πάνε στις βιομηχανικές χώρες Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Δεν μπορούν αυτά όλα να αποκαλυφθούν. Η απάντηση είναι όχι. Για να είμαι ειλικρινής, τα στοιχεία για την διαφυγή αν θέλετε για το πόσα χρήματα φεύγουν από την Αφρική. Τα δεδομένα αυτά είναι πολύ πιο σαφή και συγκεκριμένα από ότι για το ποια είναι τα εισερχόμενα στην Ευρώπη ή στη Φορή Αμερική. Τώρα πώς φεύγει φεύγουν τα χρήματα αυτά σε μετρητά ή όχι. Όχι. Γίνονται ε, ε, με άλλους τρόπους υπερβολική αύξηση των τιμών εισαγωγών ψεύτικη προφανώς και μείωση των τιμών ε, εισαγωγών και τα λοιπά. Και όπως είπε και η Ειρήν, ακριβώς αυτό το εμπορικό κομμάτι α, ε, είναι που δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα. Αποκρύπτονται δηλαδή η πραγματικότητα και πραγματικές τιμές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σαρτζεντίνη για αυτά που είπε. Τώρα, η, ιδιαίτερα για τα δημόσια μητρώα. Ναι λοιπόν, αυτό θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη αν θέλουμε να περιορίσουμε κάπως τα ποσά που διαφεύγουν από την Αφρικανική Ήπειρο. Θα μπορούσε επίσης να επεκταθεί περαιτέρω ο νόμος Ντοτ Frank. Θα πρέπει να κάνουμε και ορισμόνε, ορισμένα πράγματα για τις επιχειρήσεις του ώστε το τέλος να έχουμε στοιχεία για την κάθε μία χώρα. Ξεκινάμε για την, με την beneficial ownership και τα σχετικά μητρώα και μετά προχωρούμε σε όλα τα άλλα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Απαντάει, λέει ο κύριος Μπροκ, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε όλους που πήρατε το λόγο. Θέλετε το λόγο? Όχι. Οφείλω να πω ότι αυτοί που βγάζουν χρήματα από την Αφρική Υπάρχουν άνθρωποι που βγάζουν χρήματα από την Βόρεια Αφρική αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που παίρνουν χρήματα από την Αφρική. Ε, ε, το θέμα πάντως είναι ότι ίσως κάποιο τρόπο μπορούμε να βρούμε για να, παρά, για να ε, δούμε τι γίνονται τα χρήματα αυτά και ακούσαμε και όλο ότι τα 50 δις είναι ένα πολύ συντηρητικό ποσό. Αυτό είναι κάτι που είναι απίστευτο. Και από εκεί και πέρα ακούμε για τράπεζες που ε, τις ε, οι οποίες διασώζονται από τα λεφτά των φορολογουμένων μας και μετά εξαγοράζονται από ύποπτα άτομα ή οργανώσεις ε, της Αφρικής. Είναι λοιπόν και προς, το, προς όφελος των πολιτών μας και των φορολογουμένων μας να κάνουμε κάτι τι εδώ. Ο κύριος Λέβας... Ε, εξοχότατε Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ. Πρόκειται για ένα σοβαρότατο θέμα για την Επιτροπή Ανάπτυξης. Η κυρία Ζολή, η πρόεδρός μας, έχει κάνει κάποιες έρευνες για τα θέματα αυτά και τότε που έκανε τις έρευνες της κυρία Ζολή είχαμε ακούσει 800 δις ε απίστευτος αριθμός. Δεν ε, έχω <laughs> έχω αμφιβολία για το ότι η έκρηξη και η ε, αύξηση αν θέλετε των ακινήτων στο Λονδίνο οφείλεται πόλης σε κονδύλια, σε χρήματα σαν και αυτά για τα οποία συζητάμε. Πολλά, μα πολλά πραγματικά από τα κίνητα που αγοράζονται στην Αγγλία γίνουν, αγοράζονται με αυτά τα χρήματα προέρχονται από τις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές. Πραγματικά Είναι αδύνατο να αδιανοητό να συνειδητοποιήσει κανείς ότι αυτά τα ε, ποσά είναι τόσο μεγάλα ε, και η δική μας βοήθεια για ανάπτυξη στις χώρες αυτές είναι κλάσμα του κλάσματος του ελάχιστου ποσοστού αυτών των χρημάτων. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε.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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE να γνωρίζουμε πόσοι φοιτούν σε σχολεία, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουμε και τι είδους εκπαίδευση λαμβάνουν, τι είδους μόρφωση και αυτό θα πρέπει να έρθει στο προσκήνιο. Αυτονόητο δε είναι ότι οι στόχοι αυτοί μετά το 2015 θα πρέπει να ε, βασίζονται και στα ανθρώπινα δικαιώματα και η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει ακρογωνία λίθο της νέας ε, ε, των νέων στόχων μετά το 2015 και του νέου πλαισίου και θα ήθελα να θέσω ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πολύ συχνά εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης η πρόσβαση σε τροφή ως ε, ε, πανανθρώπινο δικαίωμα. Υπάρχουν πολυεθνικές στην Αφρική όπως άλλωστε συζητήσαμε μόλις προηγουμένως ε, οι οποίες ε, ε, προέρχονται από τις χώρες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οποίες ουσιαστικά ε, έχουν χωροκατακτητικές ε, ε, δραστηριότητες είτε για εκμετάλλευση της γης είτε για βιοκαύσιμα. Και ακούσαμε και τα έχουμε παρουσιάσει και εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης τις εκθέσεις από οργανισμούς όπως το ΦΑΟ, τον Οργανισμό για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία, και ε, βάσει των συστάσεών τους για να μπορέσουμε να θρέψουμε τον κόσμο θα πρέπει να υπάρχει βιώσιμη βιολογική καλλιέργεια και να προσπαθήσουμε να διαφυλάξουμε την ε, ελεύθερη χρήση τοπικών ποικιλιών σπόρων. το θέμα της πρόσβασης ε, του τοπικού πληθυσμού στη γη θα πρέπει να διαφυλαχθεί και θα πρέπει να ε, διασώσουμε από ε, τις κοινότητες αυτές από αυτές τις χωροκατακτητικές πολιτικές εφόσον τους δώσουμε δικαιώματα ίδιας εκμετάλλευσης της γης. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χωροταξία η οποία σχετίζεται και με καταστροφές όπως για παράδειγμα πλημμύρες. Η επιρροή των πλημμυρών ορισμένες φορές ε, σχετίζονται ε, με την έλλειψη χωροταξίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να διασφυλάξουμε και τους πόρους που έχουν αυτές οι μικρές κοινότητες και να προστατεύσουμε και τις μικρές περιοχές ε, του κόσμου που έχουν μείνει, τις λίγες περιοχές του κόσμου, συγγνώμη, που έχουν μείνει χωρίς οδικά δίκτυα. Ένα θέμα το οποίο ανακύπτει ως πρόκληση είναι οι απειλές οι οποίες προέρχονται από ε, συμφωνίες επενδύσεων και εμπορίου. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, θέτει η Επιτροπή μας σε όλες τις πολιτικές. Γνωρίζουμε ότι εμείς αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε δύο συμφωνίες ελευθερου εμπορίου και φυσικά θα έρθουν και αρκετές στη συνέχεια. Και όταν γίνεται συζήτηση για επενδυτικές συμφωνίες, αυτό το οποίο θα πρέπει να εξορθολογήσουμε είναι η ρήτρα για την επίλυση διαφορών ε, των επενδυτών για την άμεση εκμετάλλευση της ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική προστατεύει εργασιακά δικαιώματα, περιβαλλοντικά δικαιώματα, ε, ανθρώπινα δικαιώματα, μπορεί να παρουσιαστεί ως ε, ε, άμεση απαλωτρίωση της περιουσίας. Αυτό φυσικά προκύπτει και από άλλες χώρες που έχουν υπογράψει αυτές τις συμφωνίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρήτρα αυτή για να ε, υποχρεωθούν χώρες να τηρήσουν ε, συμφωνίες οι οποίες είναι αντίθετες στους στόχους της χιλιετίας. Ε, προηγουμένως συζητήσαμε τη χρηστή διακυβέρνηση, τη λογοδοσία, το κράτος δικαίου. Η διαφάνεια δεν θα πρέπει να είναι απλώς ε, αυτός σκοπός για τις κυβερνήσεις, αλλά θα πρέπει να υπερβαίνει ε, το θέμα αυτό και να είναι και στόχος των επιχειρήσεων. Ωραίο να πηγαίνουμε και να κατηγορούμε τις κυβερνήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες ότι ε, είναι διεφθαρμένες ή ότι δεν υπάρχει διαφάνεια ή ότι υπάρχει ροή χρημάτων τους ε, σε τράπεζες ε, στην Ελβετία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε φορολογικούς παραδείσους, αλλά οι πρακτικές αυτές ενθαρρύνονται και ξεκινούν από ευρωπαϊκές αλλά και άλλες πολυεθνικές. Επομένως, Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για πλήρη διαφάνεια ε, εκθέσεις ε, ε, και καταπολέμηση όλων όσων επιτρέπουν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα, νομιμοποίηση παρανόμων εσόδων, φορολογική παράδοση και ούτω καθεξής. Και φυσικά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τους στόχους της χιλιετίας από πλευράς ανάπτυξης χωρίς να ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε αυτό το 0,7% ε, και ε, το 0,15% και τις δυνατότητες να φτάσουμε στο 0,20% για το εθνικό καθάριστο εισόδημα, το οποίο θα επικεντρωθεί κυρίως στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. να πούμε ε, και κάτι θετικό, ο ιδιωτικός χρηματοπιστωτικός τομέας συνεισφέρει και σε αυτή την περίπτωση και αυτό το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, η συνεισφορά αυτή θα μπορούσε να ε, προέρθει και από το φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό, ολοκληρώνω κύριε Ντέβα, η αλλαγή του κλίματος αποτελεί όλο ένα και περισσότερο ένα μοχλό και εχθρό τους ε, επίτευξης του στόχου των, ε, της χιλιετίας. Δυσχεραίνει πολλές χώρες, δεν μπορούν να είναι λειτουργικές, ε, δεν έχουμε μόνο πρόσφυγες λόγω κλιματικών αλλαγών αλλά και για άλλους λόγους και αυτό δυστυχώς ε, θα αρχίσει να αυξάνεται ως φαινόμενο και θα είναι ε, ε, μια επονίδιστη προοπτική. Θα πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε πολύ περισσότερο πράγματα για τους φτωχότερους και τους πιο περιθεροποιημένου ανά τον κόσμο και φυσικά θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι κάποιοι από τους φτωχότερους βρίσκονται στην Ινδία, στην υποσαχάρια Αφρική. Δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τον αναπτυσσόμενο ε, κόσμο και τον αναπτυγμένο κόσμο, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε και τις φτωχότερες και πιο περιθωριοποιημένες περιοχές, κυρίως σε πιο αδύναμες χώρες. Αυτό σημαίνει φυσικά ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, ε, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ε, στόχος μείωσης κατά 50% των εκπομπών και φυσικά όπως ε, υπενθυμίζουμε στα ψηφίσματά μας θα πρέπει να υπάρχει μείωση των εκπομπών κατά 95% σε σχέση με τα ποσοστά του 1990 και μας λέγεται ότι υπάρχουν κάποιες καλές πιθανότητες να επιτύχουμε τους στόχους της υπερθέρμανσης και να μην υπάρχει αύξηση άνω των 2 βαθμών Κελσίου. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι έχουμε και άλλα θέματα ε, στην ε, γνωμοδότηση. Όπως είπατε, οι τροπολογίες είναι για του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου. Επομένως, ε, θα έχουμε και την ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα με λίγη αγάπη και να βοηθήσουμε ίσως όλες αυτές τις χώρες για τους οποίους η επίτευξη των στόχων της γενετίας θα αλλάξει πραγματικά την καθημερινότητα των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρσένη. Έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Υπάρχει όμως εδώ εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να ζητήσω λοιπόν από την κυρία Κριστίν Τιμπέρ να λάβει το λόγο για να μας πει δύο λόγια για το πώς βλέπει τους στόχους της ηλικίας και τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και δεν ξέρω και το όνομα του εκπροσώπου της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτή την έγκαιρη έναρξη των εργασιών. Εμεί θα αρχίσουμε αύριο με τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Επομένως είναι πολύ επίκαιρη η όλη διαδικασία. Επικροτούμε φυσικά το σχέδιο γνωμοδότησης και το σημείο στο οποίο εστιάζεται την επίτευξη των στόχων της ηλικία και το τι θα γίνει με την αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015. Ενδιαφέρει την τρέχουσα σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και θα απασχολήσει και την επόμενη. Ε, είχαμε το ψήφισμα πέρσι στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου στο οποίο προέδρευσα και ε, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα ε, επιτύχουμε τους στόχους της χιλιετίας, θα επικεντρωθούμε στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, για τους, ε, την αναπτυξιακή ατζέντα και επίσης συζητήσαμε και τη χρηματοδότηση πέρσι και θα ασχοληθούμε και με άλλες πηγές χρηματοδότησης που μπορούμε να έχουμε για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας και για την ατζέντα μετά το 2015. Για την ατζέντα μετά το 2015 νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη συνοχή στα όσα αναφέρονται στο σχέδιο γνωμοδότησης. Ε, θέλουμε να έχουμε ένα παγκόσμιο θεματολόγιο το οποίο θα απευθύνεται σε όλους και θα αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις και σαφώς θέλουμε να ε, δούμε τι επιτυχημένα στοιχεία είχαμε στις στόχους της χιλιετίας αλλά και πού υπήρχαν κενά. Το γεγονός ότι οι χώρες οι οποίες έχουν ε, ε, ενοπλή σύραξη και τους έχει επηρεάσει αυτό δεν μπορούν να επιτύχουν τους στόχους της χιλιετίας και θέλουμε να εργαστούμε σε αυτό το πλαίσιο να επικεντρωθούμε στην εκρίζωση της φτώχειας και στη βιώσιμη ανάπτυξη και φυσικά να δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε μια ειρηνική και σταθερή κοινωνία βιώσιμη και θέματα όπως για παράδειγμα η χρηστή διακυβέρνηση, η διαφάνεια, δημοκρατική θεσμή και κράτος δικαίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό φυσικά και σίγουρα θέλουμε να έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα να διέπουν όλο το θεματολόγιο. Επίσης θέματα φύλου, ισότητα φύλων, ε, ενδυνάμωση των γυναικών, ε, το να μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που υπάρχουν σήμερα οι γυναίκες και τα νέα κορίτσια, ε, τα οποία υπάρχουν σήμερα αλλά πρέπει να τα αναπτύξουμε λίγο περαιτέρω. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι σίγουρα όλα αυτά θα αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες για την επόμενη συνόδο των ε, Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτά μέχρι στιγμή να σα υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τρόπου... Ζητά συγγνώμη, Πρόεδρος. Όχι, δεν θέλετε το λόγο. Ωραία, λοιπόν, η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι 13 Φεβρουαρίου 5 το απόγευμα και η ψηφοφορία θα γίνει στις 3 Μαρτίου. Εάν δεν υπάρχουν από τα διάφορα κάποιοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να λάβουν το λόγο, όχι, ούτε εγώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ όλους για την παρουσία σας, για τη συνεισφορά σας. Καλό απόγευμα. Ο Πρόεδρος γενικά ευχαριστεί και τους διερμηνείς και εμείς ευχαριστούμε. Σας ενημερώνω ότι η επόμενή μας συνεδρία θα γίνει στις 3 Μαρτίου 2014 από τις 3 έως τις 6.30. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.